Αγαπητοί συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για τον κανονισμό για τον υδράργυρο. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη η σημερινή συνεδρίαση για αξιολόγηση του σχεδίου έκθεσης του εισηγητή του κυρίου ΕΚ. Του δίνω λοιπόν το λόγο για να μας εξηγήσει τη θέση του. Και κατόπιν θα έχουμε τον πρώτο γύρο παρατηρήσεων των σκιωδών εισηγητών. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη δεκαετία του 1950 στην Ιαπωνική πόλη Μιναμάτα βρέθηκαν βαρύτατες και μη επιστρεπτές βλάβες του νευρικού συστήματος και ονομάστηκε νόσος μιναμάτα που διασυνδέθηκε με τον υδράργυρο που προήλθαν από χημικό εργοστάσιο που τα απόβλητά του στην θάλασσα. 10.000 υπέστησαν σοβαρέ ζημιέ, 3.000 απεβίωσαν. Ο υδάργυρο είναι μεταξύ των 10 πλέον επικίνδυνων χημικών ουσιών στον πλανήτη μας. Πρόκειται για βαρύ μέταλλο και από τη στιγμή που θα απελευθερωθεί στην ε, φύση μπορεί να μεταδοθεί παντού με ε, αέρια μορφή προέρχεται από βιομηχανίες σε ύδατα, θάλασσες, όπου αποτίθεται σε μικροοργανισμούς και φυτά και ακολουθώντας την τροφική αλυσίδα φτάνει μέχρι τον άνθρωπο. Ο υδράγυρος μπορεί να προκαλέσει βαριές ζημιές της υγείας, βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος, του θηρεοειδούς, του ανοσοποιητικού συστήματος, των ματιών, των ούλων και του δέρματος. Τα θύματα μπορούν να υποστούν ε, σοβαρά προβλήματα μνήμης και άλλων νευρικών και άλλες επαθήσεις των νεύρων. Ιδιαίτερα βαριά θίγονται τα έμβρια και βρέφη, διότι το νευρικό σύστημα αντιδρά πολύ έντονα στον υδράγυρο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έως τώρα δεν έχει μπορέσει να θεσπίσει ασφαλές όριο για, την, για τον υδράργυρο πρόσληψης δηλαδή από τον άνθρωπο. Συχνά χρησιμοποιείται και σε χρυσορυχία και καταλήγει σε ύδατα ή και στον ατμοσφαιρικό αέρα. Επίσης κατά την κατασκευή τσιμέντου αλλά και σε ανθρακορυχία. Επίσης στην, ε, στην ανακύκλωση προϊόντων ή ως υποπροϊόν από την ε, ε, επεξεργασία κασίτερου. Ο υδράγυρος χρησιμοποιείται σε συσσωρευτές, σε λαμπτήρες, σε βιομηχανικές διαδικασίες παραγωγής. Χρησιμοποιείται επίσης και στα μείγματα που χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι για την πλήρωση κενών των οδόντων. Σε έκθεση του 2017 αναφέρεται ότι η μεγαλύτερη ζήτηση σημειώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 75 τόνοι τον χρόνο για σφραγίσματα δοντιών. Ακόμα δε και τόποι παραγωγής του υδαργύρου που δεν χρησιμοποιούνται πλέον αλλά δεν έχουν καθαριστεί αποτελούν πολύ μεγάλη πηγή κινδύνου για ανθρώπους και ζώα. Το 2013, λόγω των κινδύνων αυτών, 140 χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών υπέγραψαν τη Συμφωνία Μιναμάτα με στόχο να μειωθεί η επιβάρυνση στο ελάχιστο από υδράργυρο του περιβάλλοντος, να παρακολουθούνται και να εποπτεύονται οι εκπομπές υδραργύρου και να καταργηθούν προϊόντα τα οποία περιέχουν υδράργυρο με τον κανονισμό 1102-2008 άνοιξε ο δρόμος για την διεθνή αυτή συμφωνία και με την επιδιωκόμενη τώρα τροποποίηση του κανονισμού θα συνεχιστεί αυτή η πορεία με πιο φιλόδοξο στόχο. Ιδίω όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη τη ω προοδευτικές βιομηχανικέ χώρες θα πρέπει να είναι εκείνες μεταξύ των συμβαλωμένων μερών που θα φροντίσουν να πληρωθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν με την Συμφωνία Μιναμάτα. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν οι δεσμεύσεις αυτές λάβει την μορφή ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έχουμε τις απαραίτητες τεχνολογίες και τεχνογνωσία, μπορούμε να παραγάγουμε, προϊόντα χωρίς υδράγυρο και αυτά να τα εξαγάγουμε. Αντί όμως καλοπιστικών προσπαθειών η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει αποφάσεις που να πηγαίνουν σε βάθος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Γι' αυτό δεν μου αρέσει αυτή η μινιμαλιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δήθεν δεν δέχονται οι κύριοι Νούνκα και Τίμερμανς την προώθηση πιο φιλόδοξων στόχων. Οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απηχούν το πνεύμα τη Συμφωνία Μιναμάτα. Θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξοι στόχοι τη πρόταση αυτή και δεν προστατεύουν επαρκώ το δημόσιο συμφέρον. Οι πολίτε τη Ευρώπη απαιτούν ένα καθαρό και ασφαλή κόσμο και για του ίδιου και για τα παιδιά του. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ζήτηση υδραργύρου ανέρχεται σε 260 έως 400 τόνους τον χρόνο. Παρόλο που προβλέπεται η μείωση και μάλιστα η σταδιακή κατάργηση της χρήσης του υδαργύρου στη βιομηχανία. Και μέχρι το 2030 αναμένεται μια ζήτηση της τάξης των 40 έως 220 τόνων τον χρόνο. Με τους αριθμούς αυτούς είναι σαφές ότι με αυτές τις μινιμαλιστικές προσεγγίσεις δεν προχωρούμε. Από την αρχή της βιομηχανικής επαναστάσεως η επιβάρυνση των επιφανειακών υδάτων ανά τον κόσμο έχει τριπλασιαστεί. Στο δε βάθος της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά 25%. Σε μια επιστημονική μελέτη διαπιστώθηκε ότι σε πολλά είδη βρόσιμων ψαριών ξεπερνιέται το όριο που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το The Arctic Monitoring Program κατέληξε το 2011 στο αποτέλεσμα ότι η επιβάρυνση με υδράργυρο ε, ορισμένων ειδών ψαριών ε, των πολικών άρκτων καθώς και των θαλασσοπουλιών έχει αυξηθεί κατά ε, το δεκαπλάσιο. Κινδυνεύει λοιπόν το περιβάλλον και η υγεία των ανθρώπων διότι λόγω της βιοσορευτικής ικανότητάς του φτάνει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Απευθύνω έκκληση λοιπόν σε εσά κύριε και κύριοι συνάδελφοι να ανταποκριθείτε στις ανάγκες προστασίας που θεσπίζουν και οι συνθήκες Ευρωπαϊκή Ενώσεως για την προστασία της υγείας. Για τον λόγο αυτό έχω καταθέσει διάφορες προτάσεις τροπολογιών. Και πρώτον, να διευρυνθεί η απαγόρευση εξαγωγής υδραργύρου και για προϊόντα που περιλαμβάνουν υδράργυρο και τα οποία απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για απόβλητα με περιεχόμενο υδράργυρο. Το πρώτο αυτό, σε, καταλήγω μάλλον σε αυτό, με το συμπέρασμα ότι όλα τα προϊόντα περιλαμβάνονται στην ε, Σύμβαση Μιναμάτα πρέπει να περιλαμβάνονται και στις ε, νομοθετικές προτάσεις της Ένωσης και να αποφευθεί η χρήση διπλών μέτρων και σταθμών Όσα δεν έχουμε στη δική μας ενιαία αγορά δεν θα πρέπει να τα πολλούμε σε άλλες τρίτες χώρες. Άλλωστε είναι αντίθετο με το πνεύμα της σύμβασης της Μιναμάτα, προϊόντα τα οποία απαγορεύεται να κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά για λόγους προστασίας της υγείας, τελικώς να εξάγονται σε τρίτες χώρες. Δεύτερο, απαγόρευση ε, εισαγωγής υδραργύρου ή μειγμάτων υδραργύρου, με ορισμένες εξαιρέσεις. Καθώς επίσης η απόρριψή τους, αυτά θα πρέπει να απαγορευτούν. Τρίτο, χρήση υδραργύρου για τα ε, σφραγίσματα δοντιών. Πρώτα να απαγορευτεί σε παιδιά και εγγύους γυναίκες και μετά σε πορεία σταδιακής κατάργησης να επιτρέπεται μονάχα χρήση σε περιπτώσεις αλλεργιών στις εναλλακτικέ επιλογές. Υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογές για τα σφραγίσματα δοντιών χωρίς υδραγιο. Ορισμένες δε χώρες μέλη έχουν απαγορεύσει απολύτως την χρήση του υδαργύρου ή έχουν αρχίσει το face out. Η χρήση υδαργύρου σε κάψουλες και η χρήση διαχωριστών, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμφανίζεται ως μια δίθεν καινοτόμος λύση. Όμως, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αυτό ήδη αποτελεί πρακτική. Τέταρτο, η χρήση υδραργύρου στην βιομηχανία, όπου παίζει το ρόλο καταλήτου ή ηλεκτρολίτου. Θα πρέπει σταδιακά να καταργηθεί, διότι ήδη υπάρχουν εναλλακτικέ μέθοδοι και χρησιμοποιούνται. Πέμπτο, σε πολλές βιομηχανικές ζώνες ο υδάργυρος καταλήγει στα υπόγεια ύδατα και έτσι μολύνονται περιοχές όπου εδράζουν βιομηχανίες. Και εκεί όπου χρησιμοποιούνται χρησιμοποιείται ο υδράγυρος πρέπει να πάψει η πρακτική αυτή. Το ότι ο υδράγυρος εξατμίζεται σε θερμοκρασία δωματίου οδηγεί στο να υπάρχουν τοπικές σοβαρές παρενέργειες από τη χρήση του υδραργύρου. Προτείνεται στις χώρες μέλη όλοι οι τόποι παραγωγής προϊόντων με υδράργυρο να καταχωριστούν σε ειδικό μητρό και να απολυμανθούν το δυνατόν συντομότερο, διότι μόνο έτσι μπορούν να μειωθούν οι κίνδυνοι για φυτά ζώα και τους γειτονικούς πληθυσμούς ανθρώπων. Το ίδιο για την απόθεση του υδαργύρου και των προϊόντων υδαργύρου που λόγω μικρού όγκου και υψηλής αξίας γίνεται αυτός αντικείμενο λαθρεμπορίου. Γι' αυτό θα πρέπει ο υδραλήρος να απολύεται μόνο σε στερεά μορφή και να αποθηκεύεται μόνο σε στερεά μορφή και όχι σε υγρή μορφή. Αυτό και για την προσωρινή αποθήκευση και για την οριστική αποθήκευση. Έβδομο, νέες διαδικασίες για την ε, παραγωγή του ή για τη χρησιμοποίησή του να απαγορευτούν, ώστε να μην ανοίξουν παράθυρα για την χρήση της ουσίας αυτής που θα υπονομεύσουν την σύμβαση της Μιναμάτα. Η παραγωγή και θέση κυκλοφορία νέων προϊόντων που θα περιέχουν υδράργυρο και νέων διαδικασιών που θα βασίζονται στον υδράργυρο θα οδηγήσουν σε αύξηση της χρήσης του υδραργύρου και των ενώσεών του και σε αύξηση των εκπομπών υδραργύρου στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες νέες διαδικασίες ή νέα προϊόντα και δραστηριότητες θα πρέπει και αυτά να απαγορευτούν. Όγδο, σύστημα αναφορών παρακολούθησης της χρήσης του υδραργύρου. Για παράδειγμα, για την απόρριψη που εξαιρούνται, για την απόρριψη του που εξαιρούνται από την νομοθεσία. Στην ε, ε, βιομηχανία που χρησιμοποιεί χλώριο και αλκαλικές ουσίες. Πρέπει λοιπόν και αυτό να απαγορευτεί με τις βέλτιστες τεχνολογικές διαδικασίες. Κυρίε και κύριοι, είμαι απολύτως πεπισμένος ότι οι τροπολογίες που προτείνω εν ώψη των αδιαμφισβήτητων κινδύνων είναι αναγκαίες και ότι όντως μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από τον υδράργυρο στην υγεία φυτών, ζώων και ανθρώπων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σκιώδης ο κ. Νταντέν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη βάση εργασίας που μας προτείνει καθώς πιστεύω πως προσφέρει νομική σαφήνεια και μια προσέγγιση ε, για τον κύκλο ζωής του υδραργύρου και τη σύμβαση της ε, Μιναμάτα. Θα πρέπει να επιλέξουμε τα σωστά όργανα για να επιτύχουμε τους ε, στόχους, αλλά και να λάβουμε φιλόδοξα και αποτελεσματικά μέσα επιτόπου, ώστε να μειώσουμε τις νοσηρές επιπτώσεις του υδραργύρου, να ακολουθήσουμε τις επιστημονικές μελέτες, αλλά και θα αναγγιηθούμε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επιχειρήσης. Γι' αυτό θα προτείνω διάφορες τροπολογίε. Ε, που θα, ε, δώσουν, θα συμπληρώσουν τις ε, τροπολογίες του εισηγητή κάποιες φορές και θα συμπληρώσουν την πρόταση της Κομισιόν, αλλά είναι και αντίθετες με τις τροπολογίες του εισηγητή κάποιες φορές. Όσον αφορά την εισαγωγή υδραργύρου, οι προτάσει τη Κομισιόν είναι φιλόδοξε και σωστέ. Ωστόσο, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τη δυνατότητα να εξάγει και να εισάγει υδράργυρο για να αποφευθούν οι ελλείψει στη βιομηχανία, αλλά και για να μην τιμωρήσει τι της εταιρείας της εις βάρος προς όφελος ε, άλλων ε, μέρων του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά τα μείγματα του υδραργύρου, και εδώ η πρόταση της Κομισιόν είναι ισορροπημένη το να απεφευχθούν η εξαγωγή με βάση τη σύμβαση με δεν θα έχει θετικέ επιπτώσει στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, στο βαθμό που οι ξένε εταιρείε θα μπορούν πάντοτε να ε, εμπορεύονται αυτά τα προϊόντα. Μόνο οι ευρωπαϊκέ εταιρείε ε, θα είναι αυτέ που θα μπορέσουν να ε, ανταγωνιστούν τι ξένε εταιρείε, όπου όμω δεν τηρούν τι ίδιε προδιαγραφέ όπω οι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Ε, όσον αφορά τον ανακυκλωμένο υδράργυρο, προτείνω την εισαγωγή ενό μήνυμου στόχου χρήση υδραργύρου που προέρχεται από την ανακύκλωση. Θεωρώ ότι για τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κανονισμό, είναι καλύτερο να έχουν προέλθει από την ανακύκλωση τρία εκτήματα, καλύτερη ανείχνευση, ε, μείωση των αποβλήτων υδραργύρου και καλύτερο επίπεδο ε, ποιότητα του υδραργύρου. Όσον αφορά τη χρήση του υδραργύρου στι διάφορε κατεργασίε, για την κατασκευή εκεί όπου υπάρχει εναλλακτική θα πρέπει να απαγορευτεί η χρήση του ψευδαργυρού. μια μεταβατική περίοδο είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις ώστε να αποσβεθεί το κόστος μετατροπής των μηχανημάτων. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια μήνυμη περίοδος όταν δεν υπάρχει εναλλακτική όπως για παράδειγμα για την παραγωγή του ε, ποτάσιου. Έπειτα, η διαδικασία χωρίς υδράριο θα πρέπει να εθαρρύνει όσον αφορά τα αμαλγάματα της οδοντιατρικής. Οι οδοντίατροι έχουν ακόμα ανάγκη από αυτά τα μείγματα, γιατί σε ορισμένε περιπτώσει είναι το μόνο μείγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, ε, θα ήθελα να προσθέσουμε τρεις τροπολογίες. Μία που αφορά την πρόληψη ε, για την ε, στοματική υγεία, όπου θα πρέπει να γίνεται πρόληψη για να μειώνονται οι τεριδόνες, να προστατευτούν έτσι τα παιδιά και πρέπει να ενισχυθεί η απόδοση των, διαχωριστικών, των διαχωριστών μάλλον αμαλγαμάτων στα ε, οδοντοιατρία. Επίσης, ε, η Κομισιόν ε, δίνει την άδεια για ανταλλαγή αποβλήτων. Κάποιες τρίτες χώρες δεν έχουν οικονομικές ε, δυνατότητες ούτε και αρκετές ποσότητες υδραργύρου, για να μην μιλήσω για τις τεχνικές δυνατότητες, για να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίζει την ε, οριστική εξάλληψη αυτών των αποβλήτων και να εξαλειφθεί έτσι ο κίνδυνο κακή διαχείριση. Όσον αφορά τα απόβλητα υδαργύρου, στηρίζω τον εισηγητή. Θα πρέπει να αποφευθεί η φύλαξη υγρού υδαργύρου, που είναι πολύ επικίνδυνη για την ε, περιβαλλοντική και ανθρώπινη υγεία. Έχουμε δυνατότητε ε, για να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε την φύλαξη των αποβλήτων σε διαφορετική μορφή. Το Ευρωπαϊκό Μητρό για την ρήψη και τη μεταφορά αποβλήτων δεν νομίζω ότι είναι το κατάλληλο όργανο, γιατί αποκλείονται οι μικρέ εγκαταστάσει και η μη βιομηχανική ε, χρήση, όπω αυτή στου οδοντιάτρου. Καλύτερα είναι να γίνεται η δήλωση από όλου του φορεί, ολόκληρη την αλυσίδα. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σα για να συζητήσουμε όλα αυτά με του υπόλοιπου κοιόδου και τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παουλούτσι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τη βάση συζήτηση και ευχαριστώ τον εισηγητή ΕΚΑ για την δουλειά του που είναι σημαντική συμβολή για την εργασία μας οι εκτιμόμενες ανάγκες για υδράργυρο στην Ευρώπη ανάμεσα στο 2025 και 2030 είναι γύρω στις 40 και 200, στους 200 τόνους ετησίως. Εγώ πιστεύω ότι στόχο μας θα πρέπει να είναι να μειώσουμε στο μήνυμο απαραίτητο ε, τη χρήση του ψευδαργύρου και του, ψευδαργύρου, του υδραργύρου και να καλύψουμε τις ανάγκες από τον υδράργιο που υπάρχει ανακυκλωμένος, να μειώσουμε τη χρήση του, του υδραργύρου αλλά και να αυξήσουμε την ανάκτησή του. 100 τόνοι το χρόνο είναι ένας ρεαλιστικός στόχος ανάκτησης. Πώς και πού μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση του, του υδραργύρου. Καταρχάς, εάν μειώσουμε τον υδράργυρο στα οδοδιατρικά αμαλγάματα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που μπορούμε άμεσα να το αντιμετωπίσουμε για να υπερασπίσουμε την υγεία των πολιτών και για να αποφύγουμε σοβαρές ε, ρηπάνσεις. Εδώ μιλάμε, ζητάμε άμεση παρέμβαση να χρησιμοποιηθεί, να απαγορευτεί η χρήση των αμαλγαμάτων ε, υδραργύρου για τις ε, εγγύουση και τα παιδιά, να και να έχουμε άμεσα διαχωριστές αμαλγάματος για να αποφευχθεί η ρήπανση της γης και των υπογείων υδάτων. Δεύτερον, για τις εξαγωγές να εφαρμοστεί ε, το, οι κανόνε βέβαια που εφαρμόζουμε ισχύουν μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα πρέπει να ισχύουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ούτε διαφορετική ηθική. Η Ευρώπη πρέπει να εξάγει τι καλέ πρακτικές και άρα οι κανόνες που ισχύουν εντό Ευρώπη θα πρέπει να ισχύουν και εκτός. Και να αποφύγουμε το παράδοξο, επειδή έχουμε εμεί εδώ κάποια μεγαλύτερε βοηθικές αρχέ, να ε, αποφύγουμε την εξαγωγή προϊόντων ε, υδραργύρου που θα μας επανέρχεται όμως ως ανακυκλωμένος υδράργυρος να σταματήσει η χρήση του υδρογύρου εκτός από εκεί όπου έχει αποδεδειγμένα ε, αποδειχτεί τη χρήσιμη χρήση του και εκεί που δεν υπάρχει εναλλακτική να πάψει να χρησιμοποιείται ε, η, χρήση του υδραργυρίου για την παραγωγή εθοξιδίου και μεθοξιδίου του νατρίου ε, και του ποτασίου. να σταματήσει η εισαγωγή προϊόντων που περιέχουν υδράργιο στις, ε, μέσα στην αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού. Εάν αναλάβουμε το σύνολο αυτών των μέτρων και αν δουλέψουμε σοβαρά για την ανάκτηση, είναι δυνατόν να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θεσπίσει. Έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες ε, αντιμετωπίσει σοβαρά το θέμα του κατά πόσο ήταν σωστό ή όχι η Ευρώπη να δεχτεί την εισαγωγή υδραργύρου ως απόβλητου. Οι ενδείξεις που μας, που φτάνουν από ένα σωρό περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι ότι στην Ευρώπη υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να υπάρξει καταργασία του υδραργύρου υπό συνθήκες που δεν υπάρχουν εκτός Ευρώπης. Και άρα και αν λάβουμε υπόψη το σύνολο της, ποιότητα ποιότητας του περιβάλλοντος θα ήταν καλό να επιτραπεί η εισαγωγή υδραργύρου προς ανακύκλωση. Και τέλος όσον αφορά τα απόβλητα στην Ευρώπη θεωρούμε πως θα πρέπει να σταματήσει η εξαίρεση ότι δηλαδή ο υδράριος μπορεί να αποθηκεύεται σε υγρή μορφή. Θα πρέπει να εισαχθεί με μάλιστα συγκεκριμένο χρονικό όριο ένα, μια δυνατότητα στερεοποίησης και έπειτα θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει και ένα μητρό που θα εγγυάται τη δυνατότητα παρακολούθησης και ανεχνευσιμότητας του αποβλήτου αυτού. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Γκέρλινγκ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο κούρεμα. Ήθελα να υποβάλω κάποιες προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον δεν με άκουσε ο Πρόεδρος. Ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι μου φαίνεται ότι η ισορροπία είναι αρκετά σωστή, ότι ξεκινούν στο σωστό σημείο. Θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ε, υπό την σύμβαση της Μιναμάτα. Θα πρέπει να προσπαθούμε να κλείσουμε κενά και να βελτιώσουμε τον τρόπο που δουλεύουμε. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι για να πετύχουμε το μέγιστο όφελος θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα θέμα παγκόσμιο και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενεργήσει εντός αυτού του παγκοσμίου πλαισίου. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πέρα από τις υποχρεώσεις της Ευρώπης ε, σύμφωνα με την Σύμβαση της ε, Μιναμάτα και πώς μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερο περιβαλλοντικό όφελος. Όσον αφορά λοιπόν ε, αυτή την πλήρη απαγόρευση εξαγωγών, κάτι που θέλει πολύ ο εισηγητής, δεν είμαι και πολύ βέβαιη. Κοιτώ την ε, μελέτη αντικτύπου της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν έχω πιστεί ότι εάν απαγορεύσουμε τις εξαγωγές δεν θα μεταφέρουμε απλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόβλημα. Φυσικά, μακροπρόθεσμα θέλουμε μηδενική χρήση υδραργύρου, αλλά ίσως είναι καλύτερα να ελέγχουμε την κατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για περιβαλλοντικούς λόγους. Δεν δέχομαι λοιπόν απαραίτητα ότι η απόλυτη απαγόρευση εξαγωγών είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Επίσης, όσον αφορά τις εισαγωγές, ο εισηγητής έχει επιλέξει ε, μία οδό που απορρίφθηκε από την μελέτη αντικτύπου. διότι φαίνεται ότι η απαγόρευση εισαγωγών θα οδηγήσει σε περισσότερη προμήθεια υδραργύρου σε αναπτυσσόμενες χώρες ε, όπου ε, μπορεί κιόλας να χρησιμοποιείται για ε, χρυσορυχία μικρής κλίμακας και μπορεί αυτή να είναι η επόμενη καταστροφή για τον πλανήτη μας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει ότι α, εμείς το απαγορεύσαμε αλλά θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα σε άλλα μέρη του κόσμου. Και όσον αφορά τα δύο αυτά θέματα, λοιπόν, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει δίκιο. Όχι ότι δεν μπορούν να γίνουν κάποιες λεπτές ρυθμίσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τη συμμόρφωση με τη Σύμβαση. Νομίζω ότι ο εισηγητής έχει δίκιο όταν ε, ζητάει σφίξιμο των ε, διατάξεων της Σύμβασης σε κάποια σημεία. Εάν δεν μπορούν να αποδειχθούν ε, περιβαλλοντικά ωφέλη, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απογορεύσουμε τη χρήση του υδράργυρου σε νέα προϊόντα, κάτι που μπορεί να γίνει ε, βαθμιαία με μια σειρά τροπολογιών. Και όσον αφορά τα, τον υδράργυρο στην οδοντογιατρική, ε, εγώ που έχω το στόμα μου γεμάτο υδράργυρο, μπορώ να σας πω ότι νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα να ε, καταργήσουμε τελείωσε την χρήση του υδραργύρου. Ξέρω ότι οι ενώσεις οδοντιάτρων ε, θέλουν να χρησιμοποιούν ε, υδράργυρο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου το αμάλγαμα υδραργύρου να είναι το καλύτερο υλικό, αλλά Ήδη υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τον εισηγητή ότι θα πρέπει η θέση εκκίνησή μα ε, να είναι μη χρήση στην οδηγιατρική και να προβλέψουμε παρεκκλήσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιατανμάκη. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι που βλέπω ότι γενικά συμφωνούμε στο θέμα αυτό. Ο υδράργυρος είναι ουσία πολύ επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία. Και γι' αυτό η κύρωση της σύμβοσης της Μιναμάτα είναι πολύ σημαντικό θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι θα πρέπει να νομοθετήσει πολύ πιο αυστηρά για τον υδράργυρο από ό,τι ε, ισχύει αυτή τη στιγμή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε πιο αυστηρούς κανόνες. Και κάποιες παρατηρήσεις για την ε, έκθεση του Στέφαν Εκ. Καταρχάς, ε, συμφωνώ με, την, ε, με τον στόχο του εισηγητή να έχουμε νομική βάση. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε τα ίδια πρότυπα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες όσον αφορά την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο. Οι τρίτες χώρες που δεν έχουν ε, την σωστή τεχνολογία για τον χειρισμό του υδραργύρου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στην Ευρώπη ε, τα επικίνδυνα απόβλητα για να γίνει σωστή επεξεργασία του, Όσον αφορά τον οδοντιατρικό υδράργυρο, δεν συμφωνώ απολύτω. θα πρέπει να μειωθεί ε, η χρήση του υδραργύρου στην οδοντιατρική και αυτό συνάδει με το πνεύμα της σύμβασης της Μιναμάτα. Η χρήση τέτοιων φλαγισμάτων ε, θα πρέπει να εγκρίνεται εφόσον είναι η μόνη δυνατή λύση σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. Ο εισηγητής έχει υποβάλει κάποιες τροπολογίες που διευκρινίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμφωνώ με την ε, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ώστε να μην χρειαζόμαστε υδράργυρο στο μέλλον και να έχουμε ε, μείωση του αριθμού των προϊόντων ε, στα οποία χρησιμοποιείται υδράργυρο στο μέλλον. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία που σχετίζεται με τον υδράργυρο και να προχωρήσουμε στην πλήρη κατάργηση της χρήσης του υδραργύρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πελόζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ακούω τους συναδέλφου, νομίζω πω μπορούμε να συμφωνήσουμε για κάποια πράγματα. Τώρα ακόμη και η Κομισιόν συμφωνεί ότι ο υδράριο είναι απειλή για την υγεία και το περιβάλλον παγκοσμίω. Έχουμε λοιπόν το καθήκον να είμαστε φιλόδοξοι ώστε να ξεφορτωθούμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά και όσο γίνεται πιο γρήγορα τον υδράριο. Η πρόταση της Κομισιόν για μένα όμως δεν προχωρά αρκετά και χαίρομαι για τη θέση του εισηγητή που τη βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό και θα καταθέσουμε και τροπολογίες όσον αφορά την εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς η Ευρώπη μπορεί να εξάγει κάποια τέτοια προϊόντα ενώ ε, τα απαγορεύει εντό της εσωτερική αγοράς. Θα πρέπει τι να μπορούμε να εξάγουμε τις ε, μπαταρίες ε, μιας χρήσης ή τις ε, φωσφορίζοντες λαμπτήρες. Δηλαδή είναι μια μικρή αγορά, μια αγορά που προστατεύει την Ευρώπη και μια αγορά όπου οι κανόνες ξεπερνούν αυτούς της εσωτερικής αγορά. Αυτό δεν είναι δυνατόν έπειτα για τη χρήση του υδράργυρου. Έχουμε την χρήση για τα οδηγητικά αμαλγάματα και μετά έχουμε το ότι αφορά το χλώριο, το θείο και τα λοιπά. Για τα οδηγητικά αμαλγάματα ξέρουμε ότι τα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο ήδη θεωρούνται επικίνδυνα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα αμαλγάματα. Πρέπει να να γυρίσουμε σελίδα. Εδώ λέει για το Δεκέμβριο 2021 ως ε, όριο. Έχουμε λοιπόν περιθώριο για να βρούμε και εναλλακτικέ. Μα δείτε, η Δανία και η Σουηδία ήδη δεν χρησιμοποιούν ε, υδράργυρο ε, στα, στον διαιτητρική. Ε, διάφορα διάφορα άλλα μείγματα ε, χρησιμοποιούν και για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Υπάρχουν εναλλακτικές. Έχω συζητήσει με τους οδοντίατρους. Είναι τόσο, ε, τόσο συνηθισμένοι να χρησιμοποιούν αυτά τα αμαλγάματα που λένε ότι είναι πανεύκολο να τα χρησιμοποιήσει. Πρέπει απλά να αλλάξει την πρακτική. Ας τους αφήσουμε λοιπόν μέχρι το 2021. Αν τους πούμε ότι το 2021 τέρμα τα, αυτά τα οδοντιατρικά αμαλγάματα εν πάση περιπτώσει σε πολύ εξαιρετικέ περιπτώσει. Ε, πρέπει να προσέξουμε όμως γιατί και στις εναλλακτικέ ή σε κάποια άλλα μείγματα δεν πρέπει να υπάρχει ούτε δυσφενόλη. Όχι, υπάρχουν διάφορα παράγωγα. Και ο ΠΟΗ λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνο σε αυτά. Άρα κανένα πρόβλημα. Εκεί που χρησιμοποιείται πολύ ο υδράριος είναι η βιομηχανία του χλωρίου γιατί εκεί ε, δεν μπορούμε, πάλι υπάρχει τεχνολογία και η εναλλακτική και πρέπει να δοθεί μια μεταβατική περίοδο και ένα επίπεδο όπου να είναι απαγορευμένο. Έπειτα για τους καταλήτες για να παράγεται το βιοντίζελ. Και εδώ υπάρχουν εναλλακτικέ ευρωπαϊκές εταιρείε που παράγουν ε, άλλα υλικά ε, όπως για να φτιάξουν μάλλον το μεθοξίδιο του νατρίου που δεν χρησιμοποιούν υδράργυρο. Μετά το θέμα της, ε, των αποβλήτων του υδραργύρου, τα αστεριά και τα υγρά απόβλητα. Η Κομισιόν να προτείνει την αποθήκευση υγρή μορφή δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει... Ε, η αδρανοποίηση, η νερτάζ. Δηλαδή δεν είναι στερεοποίηση, αλλά γίνεται αδρανοποίηση του υλικού. Θα πρέπει να υποχρεωθούν όλες οι χώρες όπου έχουν στερεά και υγρά απόβλητα να τα αδρανοποιήσουν και να τα βάλουν σε μια μεταβατική αποθήκη. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν αυτή τη τεχνολογία. Αλλά Υπάρχουν γερμανικές εταιρείες που αυτή τη στιγμή κάνουν και κινητή αδρανοποίηση, δηλαδή μεταφέρεται η τεχνολογία έτσι ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να μετακινούνται στην κάθε χώρα για να κάνουν αδρανοποίηση. Αν αρχίσουμε να δεχόμαστε τώρα την εισαγωγή αποβλήτων, ξέρετε όσο εισάγουμε απόβλητα τόσο θα χάνουμε και την ανιχνευσιμότητα και έχουμε παραδείγματα όπου έγιναν διάφορα, διάφορα μπερδέματα. Ε, λοιπόν, υπάρχει τεχνολογία για την αδερμοποίηση και την αποθήκευση και δύο λόγια για την οριστική αποθήκευση, γιατί υπάρχει μεταβατική και η οριστική. Λοιπόν, με την εμπειρία που έχουμε, όταν είδαμε τι γινόταν στη Γερμανία, στο Καμίν, στο Στρασβούργο, ε, ο κάθε φορά που αποθηκεύουμε σε μεγάλο βάθος, είτε στην, ε, στα ορυχεία όπου κάποια στιγμή κατέπεσε η οροφή ή στην ορυχία του ΣΕΡ όπου πλημμύρισε η συγκεκριμένη ε, χωματερή του ΑΣ στην Γερμανία. Όχι αποθήκευση λοιπόν σε μεγάλο βάθος, στην επιφάνεια για να μπορούμε να παρέμβουμε αν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτά τα απόβλητα διαρκώς σωρεύονται και δεν καταστρέφονται. Είναι σαν τα διενεργά απόβλητα. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει επάπειρον εσαι να μπορούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται. Και ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή γιατί έχει κάνει πολύ καλές προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Ντορνανό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η μόλυνση χιλιάδων ανθρώπων ανάμεσα το 1932 και το 1966 στην Ιαπωνία, που είναι γνωστή ως ασθένεια της Μιναμάτα, αποτελεί τρανό παράδειγμα, τραγικό αλλά και διάσημο για την ακραία νοσηρότητα αυτή Τη τη ουσία στην υγεία. Τη βρίσκουμε σήμερα στα ψάρια αλλά και σε αντικείμενα που κατασκευάζονται όπω τα θερμόμετρα, οι ε, ε, λαμπτήρες και τα οδοντιδικά μαργάματα. Αυτό ήδη υπόθηκε. Επίση χρησιμοποιείται στη βιομηχανία σε διάφορε διαδικασίε εξόριξη χρυσού. Τον Οκτώβριο του 2013, 139 χώρε, μεταξύ των οποίων 26 ευρωπαϊκέ χώρε, εκτό από τη Λετωνία και την Πορτογαλία, υπέγραψαν στην Ιαπωνία τη σύμβαση τη Μιναμάτα για τον υδράργυρο. Πρόκειται για σημαντική πρόοδο γιατί είναι διεθνής, διεθνές το πεδίο εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το α και το ω σε αυτή την υπόθεση, γι' αυτό και η προσφυγή στις κατεξουσιοδότηση και στις εφαρμοστικές πράξεις θα πρέπει να είναι ο κανόνας αλλά η εξαίρεση. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την ε, κυρίαρχη θέληση της, της και της Πορτογαλίας, αλλά να καλέσουμε τις χώρες αυτές σε έναν επικοδομητικό διάλογο, ώστε να υπογράψουν και αυτές τη σύμβαση της Μιναμάτα. Η Κομισιόν θα πρέπει να αποκλείει τα κράτη από αποφάσεις που έχουν να κάνουν με περιορισμό των εξαγωγών ή των εισαγωγών το ίδιο. Όσον αφορά την αδειοδότηση για νέα προϊόντα, για νέες διαδικασίες παραγωγής που περιέχουν υδράργυρο, ή για το θέμα της τροποποίηση των παραρτημάτων, για την εφαρμογή της σύμβασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες φορές ξεχνά ότι τα κάτι μέλη είναι κυρίαρχα και αυτόνομα έχουν αναλάβει διεθνεί δεσμεύσει, μπορεί επίση να υποβάλει στη γραμματεία αυτή τη σύμβαση μια ανέκθεση το όνομά της, αλλά όχι στο όνομα των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Miss Ευχαριστώ, η κυρία Αγιούζο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ επίσης ε, τον εισηγητή και τους Σκιώδης. Ε, η πρόταση αυτή... Ναι, αυτό είναι είναι η σύμβαση, είναι, η της Μιαμάτα είναι πολύ σημαντική και επίσης είναι απογοητευτική η πρόταση της Κομισιόν γιατί ε, σημειώνει την ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ε, είναι απογοητευτική και από διεθνή άποψη και το είπε και ο σύμβουλος, το Συμβούλιο μάλλον γιατί ε, δεν τηρεί ούτε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε με τη σύμβαση της Μιαμάτα Ωστόσο, Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για τη συνέταξη. Καλή έκθεση και ε, τονίζει αυτά τα σημαντικά ε, ε, σφάλματα, για παράδειγμα όσον αφορά τον περιορισμό χρήσης που περιλαμβάνεται στο τρίτο παράρτημα και συγκεκριμένα για την ε, παραγωγή εθοξιδίου, μεθοξιδίου του νατρίου και του ποτασίου. Δέχεται ότι χρησιμοποιείται ο υδράργυρος και ορίζει πολύ περιορισμένες μεταβατικές περιόδους για να πάψει η χρήση του ε, υδραργύρου, όπως λέει εξάλλου και η Σύμβαση της Μιναμάτα. Τώρα, όσον αφορά την, ε, τα απόβλητα υδραργύρου, έχουμε να, έχω να πω τα εξή. Καταρχά, είναι αδιανόητο η Κομισιόν να επιτρέπει την αποθήκευση, τη μόνιμη μάλλον αποθήκευση σε υγρή μορφή, όπω είπε και η κυρία Ριβασί, αντίθετα με το γενικό κανόνα για τα απόβλητα. Ένα υγρό απόβλητο είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κανεί και να το ελέγξει και δεν είναι σταθερό γιατί μπορεί να εξατμιστεί. Είναι ένα από του μεγαλύτερου κινδύνου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τον υδράριο. Σύμφωνα με τη Σύμβαση τη Βασιλεία, στην οποία παραπέμπει και η Σύμβαση τη Μιναμάτα, τα απόβλητα υδραργύρου ή τα μείγματα υδραργύρου θα πρέπει να στερεοποιηθούν πριν ε, εξαλειφθούν. Επίσης υποχρεώνει να αποθηκεύονται μόνο τα απόβλητα που έχουν περάσει από κατεργασία. Δηλαδή η Κομισιόν επιλέγει την λιγότερο αυστηρή ε, ε, δυνατότητα που υπάρχει. Εξάλλου επιτρέπει μόνο την υπόγεια μόνιμη αποθηκεύση χωρίς κανένα είδος αξιολόγησης. Εγώ πιστεύω ότι ο υδράργυρος η εμαθήκευσή του μάλλον σε υπόγειους χώρους είναι υποχρεωτικός μόνο για τα ραδιενεργά απόβλητα, λόγω της ραδιενέργειας που εκπέμπουν. Ενώ στην περίπτωση του υδραργύρου δεν υπάρχει ε, ραδιενέργεια και γι' αυτό είναι καλύτερη η επιφανειακή αποθήκευση, γιατί έτσι ελέγχεται καλύτερα και αποφύγεται η, ε, στα υπόγεια ύδατα και μπορεί κανείς να παρέμβει ε, γρήγορα και εύκολα σε περίπτωση επίγουσας ανάγκης. Είναι μια επιλογή που πάντως πρέπει να μελετηθεί καλύτερα. Ε, έπειτα, η Επιτροπή απαιτεί ή μάλλον μας προτείνει μία στάνταρ αποθήκευση, δηλαδή η, τα χωρίς όμως καμιά δικαιολογία. Σε καμία από τις σελίδες της μακροσκελούς πρότασης δεν υποδεικνύει καμία εναλλακτική αποθήκευση σε επιφανειακή κτλ. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη σε όλες αυτές τις σελίδες. Η ταλατορυχία είναι ίσως ένας από τους πιο εύκολους τρόπους αποθήκευσης αποβλήτων, όμως δεν προσφέρει καμία ασφάλεια και επιπλέον υπάρχει δίσδυση νερού πολύ επικίνδυνη γιατί το αλάτι είναι εξαιρετικά διαβρωτικό. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να μελετήσει καλύτερα τις επιλογές και εν τέλει ναι, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Μας προτείνει μια εναρμόνιση προς τα, προς τα κάτω. Υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν τεχνικές που μπορούν να τα λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ ζω 100 χιλιόμετρα από το μεγαλύτερο ορυχείο υδραργύρου στον κόσμο που είναι, ε, λειτουργεί από την εποχή των Φινίκων και υπάρχουν τεχνικοί που εργάζονται όλη τους τη ζωή με τον υδράργυρο και ποτέ δεν υπήρξε εκεί ατύχημα και έχει μάλιστα καταθέσει την ευρεσιτεχνία για την επιλογή της κατεργασίας και της επεξεργασία των αποβλήτων. υπάρχουν πολύ καλές επιλογές, πρέπει να τις μελετήσει η Κομισιόν. Εγώ θα καταθέσω και θα τη συζητήσω και με τους υπόλοιπους ισκιώδεις βεβαίως. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, ο κύριος Φλόρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κανείς νομίζω δεν θα αρνηθεί το ότι ο υδράγυρος είναι από τις πιο επικίνδυνες τοξικές ουσίες που γνωρίζουμε. Ωστόσο θέλω να επισημάνω ότι τα τελευταία 20 χρόνια κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει περί υδραργύρου. Εσείς ήσασταν τόσο νέος που δεν τα γνωρίζετε. Έχουμε συζητήσει μέχρι λιποθυμίας το θέμα αυτό. Έχουμε, έχουμε ε, ψηφίσει νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν εφαρμόζονται. Δεν χρησιμοποιείται καν ο υδράγυρος πλέον σε σφαγίσματα δοντιών. Πρόκειται μόνο για την εξαγωγή. Βεβαίως, ως απόβλητο βάλτε ανθρώπους στα σύνορα να προσέχουν να μην συμβαίνει αυτό. Τώρα αυτή η γενική απαγόρευση υδραργύρου εμένα δεν θα μου άρεσε διότι πρέπει πολύ περισσότερο να εξεταστεί πόσο ασφαλής είναι η χρήση του. Υπάρχουν δωδεκάδες χρήσεις υδραργύρου που πραγματικά δεν έχουν εναλλακτική επιλογή και αυτό που πρέπει, στο οποίο πρέπει να εγγύψει κανείς είναι η ασφάλεια της χρήσης του υλικού αυτού. Βεβαίως, αν κάποιος ή κάποιοι πετούν τα πράγματα αυτά τα σκουπίδια, ασφαλώς αυτό αποτελεί αμέλεια. Όμως, εάν μια βιομηχανία που παράγει προϊόντα, για παράδειγμα, ζανιοκτώνα, δεν μπορεί να, και χρησιμοποιεί το δεν μπορεί κανείς να τη βάζει εμπόδια στο δρόμο της. Πάμε τώρα να επινοήσουμε νέα μέτρα προστασίας των φυτών. Ένα όμως προϊόν το οποίο είναι πρόδρομος αυτών των ε, ε, ουσιών και επομένως χρειάζεται, πάμε να το απαγορεύσουμε. Λοιπόν, πολιτική μονάχα με απαγορεύσεις είναι υπεραπλούστευση. Χρειάζεται να εξετάσουμε επιμέρους ρυθμίσεις, να εξετάσουμε ακριβώς πού σημειώνεται ο κίνδυνος Ήδη πριν από 20 χρόνια απαγορεύσαμε τα θερμόμετρα πυρετού με ε, υδράλιο. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι ορισμένες χρήσεις μπορεί να ανασφαλίσει και πρέπει να επιτρέπονται για να δώσουμε στην βιομηχανία και τη δυνατότητα να επινοήσει καινοτόμα προϊόντα. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε θα πρέπει να δούμε στο μέλλον τι, ε, πού θα έχουμε κάποιες ευκαιρίες. Ασφαλώς και θα υποβάλω τροπολογίες, υπάρχουν και κάποια κενά. Έχω να πω κάτι ακόμη ήδη ως πρόεδρος της Επιτροπής για την οδηγία Ριτς είχα σπάσει τα μούτρα μου με 2.000 τροπολογίες. Και οι μισές από αυτές, αν ήταν σαν αυτές που λες εσύ, δεν θα είχε φτάσει ο Ιδάγιος ποτέ να δει το φως του κόσμου. Το ζήτημα είναι λοιπόν ποια είναι η χρήση, πώς γίνεται η χρήση του υδαργύρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαγορεύεται απολύτως η χρήση του και καλώς. Όμως σε άλλες περιπτώσεις χρειάζονται βεβαίως ρήτρε ή ρυθμίσεις προστασίας και αυτών που χρησιμοποιούν τον υδράγυρο στην παραγωγή προϊόντων. Εντάξει, ας γίνει σε δύο-τρία χρόνια μια επανεξέταση. Όμως, δεν μπορείτε να απαγορεύσετε τα πάντα στη βιομηχανία, διότι σιγά σιγά θα πρέπει να σκεφτόμαστε πού θα βρίσκουν απασχόληση οι άνθρωποι. Ευχαριστώ κύριε Φλόρεντς. Ο κύριος Μικολάσικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ στο θέμα αυτό. Εξέτασα προσεκτικά το θέμα και έχω διαπιστώσει τα εξής. διότι ζητώ να υιοθετήσουμε ρεαλιστική προσέγγιση. κατά την ε, αξιολόγηση των ε, διαφόρων λύσεων. Λέγεται να απαγορεύσουμε τον υδράργυρο όπου αυτό είναι δυνατόν. Ε, συμφωνώ και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες λύσεις. και όπου είναι δυνατόν, όπου υπάρχει εναλλακτική λύση, θα πρέπει να αντικαθίσταται ο ψευδάργυρος. Και θα πρέπει να αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις και εναλλακτικά υλικά. Για παράδειγμα, Αναφέρθηκαν ε, διάφορες ε, ουσίες ε, που δρούν ως καταλύτες ή ηλεκτρόδια και πρέπει να πω ότι έχουμε διάφορες διαδικασίες παραγωγής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αληθεύει αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες αυτές πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μεταβατικές περιόδους για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να απαγορέψουμε την χρήση του υδραργύρου. σε περιπτώσεις άλλων ουσιών ε, ακολουθήσαμε πολύ ισορροπημένη προσέγγιση σας καλώ λοιπόν και εδώ να προσαρμόσουμε ανάλογα τις μεταβατικές περιόδους. Θα ήθελα δηλαδή ως προθεσμία να έχουμε τον ε, Δεκέμβριο 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σλίνς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρκετοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην απαγόρευση εξαγωγών. Στον ισχύοντα κανονισμό προβλέπονται παρεκκλήσεις για την έρευνα και για γιατρικούς σκοπούς. Στην ε, νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η παρέκκληση από την απαγόρευση εξαγωγών προβλέπεται μόνο για την έρευνα. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την παρέκκληση για γιατρικούς σκοπούς, τι γίνεται. Για τα ομοιοπαθητικά φάρμακα χρειαζόμαστε ε, τον υδράργυρο σε ελάχιστες ποσότητες. Είναι απαραίτητη η ουσία αυτή στην ομοιοπαθητική. Ε, έχει να προτείνει κάποια λύση για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Κροστέτ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη γιατί α, ήδη υπόθηκαν αρκετά πράγματα. Πρέπει να πω ότι είμαι σύμφωνη με την γνώμη των υπολείπων ότι όντω ο υδράργυρο είναι κίνδυνο για την υγεία και για το περιβάλλον. Ωστόσο, πιστεύω πω η θέση του εισηγητή είναι εξαιρετικά σκληρή σε σχέση με τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, με έβρισκε πιο σύμφωνη. Υπάρχουν διάφορε τροπολογίε του εισηγητή που με ανησυχούν κάπω διότι ζητά μια πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών ε, υδραργύρου καθώς και της ε, παραγωγής και του εμπορίου προϊόντων που περιέχουν ε, υδραργύρο όμως ο προηγούμενος συνάδελφος το είπε μόλις ότι θα ήταν τέτοιοι κανόνες αντιπαραγωγικοί. Γιατί, Γιατί στο τομέα της φαρμακευτικής χρησιμοποιείται ακόμα ο υδράργυρος ειδικά στα ομοιοπαθητικά φάρμακα και στα εμβόλια όπου χρησιμοποιούνται παράγωγα υδραργύρου και αυτά τα ε, παράγωγα είναι εγκεκριμένα από τις αρχές των φαρμάκων και ε, αυτή τη στιγμή φέρνουν ωφέλη. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε. Αν πρέπει κάποια στιγμή να απαγορευτεί η χρήση του υδραργύρου, θα πρέπει να έχουμε και απαραίτητε μεταβατικέ περιόδου για να βρεθούν οι εναλλακτικέ. Γιατί για την ώρα σε ορισμένου τομεί δεν υπάρχουν. Αυτά είχα να πω. Γιατί όταν είμαστε πολύ αυστηροί και άκαμπτοι, μπορεί να κάνουμε λάθος. Ναι, λοιπόν, στις, ε, στους περιορισμούς ε, της χρήσης του υδραργύρου, να, ναι, να φτάσουμε στην απαγόρευσή του, αλλά με μεγάλη προσοχή. Σε ορισμένους τομείς χρειάζονται ακόμα τα παράγωγα του. Υδραργύρου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκροστέτ. Και τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, κυρία Winning. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Στην απάντησή μου θα επικεντρωθώ στο γενικό πλαίσιο της πρότασής μας ε, και θα απαντήσω σε κάποια από τα σημεία κλειδιά που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Σας ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις οι οποίες ε, νομίζουν, νομίζω συμβάλλουν θετικά στην συζήτηση που μας περιμένει και σε διοργανικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, από τις ε, πρώτες χώρες όσον αφορά την πολιτική για τον υδράργυρο. Έχουμε μειώσει τη χρήση του κατά 80% και έχουμε περιορίσει τη χρήση του σε προϊόντα και διαδικασίες. Ε, με τις νομοθεσίες REACH και την σχετική οδηγία. θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το 40 με 80% που ε, απομένει ως κατάλοιπο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από άλλα μέρη, της, από άλλα μέρη του κόσμου. Περιβαλλοντική διπλωματία αντιπροσωπεύει η σύμβαση της ε, Μιναμάτα και βασίζεται στο κοινοτικό κεκτημένο θα μειώσει ριζικά τις ε, τις ποσότητες ε, υδρατηγύρου σε όλο τον κόσμο και επίσης ε, θα δημιουργήσει συνθήκες ίσου ανταγωνισμού καθότι όλες οι μεγάλες οικονομίες θα πρέπει να εφαρμόζουν παρομοίες απαιτήσει και αυτό θα ευνοήσει και την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την καινοτομία που αναζητά εναλλακτικές λύσεις. Ενώ λοιπόν θέλουμε να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας ε, για την υγεία των πολιτών και για το περιβάλλον, ευθυγραμμίζουμε και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την Σύμβαση. Επίσης, απαγορεύουμε την ε, νέα χρήση υδραργύρου σε προϊόντα ή βιομηχανικές διαδικασίες που να μην ωφελούν την υγεία ή το περιβάλλον και θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου και ε, ε, επιβεβαιώνει την ηγετική μας θέση σε όλο τον κόσμο όσον αφορά την μείωση ε, των επιπέδων ιτεραγύρου. Να απαντήσω όσον αφορά τα ιατρικά αμαλγάματα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το να προχωρήσουμε πέρα από τις απαιτήσεις της σύμβασης και προτείναμε να είναι υποχρεωτικός ο διαχωρισμός των αμαργαμάτων για να μειώσουμε την ε, μόλυνση του νερού και επίσης να χρησιμοποιούνται τρόποι ώστε να προστατεύονται οι οδοντίατροι και οι ασθενείς από ε, τις ε, επιπτώσεις του υδραγύρου. Δεν έχουμε απαγορεύσει όμως απολύτως τον οδοντιατρικό υδράργυρο. Επίσης αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση ότι διάφορα κράτη-μέλη έχουν διάφορα προγράμματα ή διάφορα μέτρα και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι καλύτερα σε θέση ε, να επιλέξουν εναλλακτικέ λύσεις. Όσον αφορά τα απόβλητα, προτείνουμε να ε, αφήσουμε ανοιχτή την ε, δυνατότητα ε, να υπάρχει δυνατότητα υπόγειας αποθήκευσης ε, των αποβλήτων ε, για να αποφύγουμε νέα σκάνδαλα εξαγωγών υδραργύρου που είδαμε τις τελευταίες δεκαετίες που ήδη έχουν βλάψει την φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν τα κράτη-μέλη επιτρέπουν μόνο αποθήκευση στερεού υδράργυρου και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν στην αγορά νέοι ε, τρόποι διάθεσης ε, των αποβλήτων. Ε, μόνο μία λύση έχει προταθεί και δεν έχει φανεί να υπάρχει κάποια ρεαλιστική λύση. Τότε θα πρέπει να αποθηκεύεται επί 10 χρόνια ο υδράργυρος μέχρι να σταθεροποιηθεί. Κάτι που θα πρέπει να συνοδεύεται από συστήματα ελέγχου και ηχνηλασιμότητας κάτι που επιβάλλει επιπλέον διοικητικό άχθος. Επίσης, όπως υπόθηκε νωρίτερα, η ε, απαγόρευση εξαγωγών υδραργύρου μπορεί να μεταφέρει την χρήση του υδραργύρου σε τρίτες χώρες όπου η έλεγχη να μην είναι ε, τόσο αυστηρή και έτσι να μην πετύχουμε ε, τους περιβαλλοντικούς μας στόχους μπορεί να περιπλέξει την λήψη μελλοντικών αποφάσεων όσον αφορά τα πρότυπα της αγοράς μας. Γι' αυτό ο καλύτερος τρόπος ε, για μας είναι να εφαρμόσουμε πρώτα την ε, σύμβαση με τους εμπορικούς μας εταίρους και κατόπιν να χρησιμοποιήσουμε τη ρήτρα αναθεώρησης της σύμβασης για να πείσουμε τους εταίρους μας να επεκτείνουν τους ε, ελέγχους των προϊόντων ε, εισάγοντας ε, στη Σύμβαση Μιναμάτα νέα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα πιο αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, Υπάρχει το θέμα των ε, ενώσεων υδραργύρου στην ε, φαρμακευτική βιομηχανία. Πιστεύουμε ότι οι παρεκκλήσεις ε, στην απαγόρευση εξαγωγών είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν ούτως ή άλλως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει παρεκκλήσεις μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία. Η χρήση του υδραργύρου στην φαρμακοβιομηχανία είναι πολύ περιορισμένη και πιστεύουμε ότι υπάρχει ε, ότι υπάρχουν επαρκείς ποσότητες ε, στον κόσμο χωρίς να απαιτούνται εξαγωγές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την ε, εισαγωγή ε, υδραργύρου, συγγνώμη. Πιστεύουμε ότι μειώνεται η ζήτηση του υδραργύρου ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων ε, για τα προϊόντα και τις ε, διαδικασίες. Ωστόσο, θα ε, συνεχίσει να υπάρχει ανάγκη εισαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον όσο οι κατάστασεις ανακύκλωσής μας δεν παράγουν επαρκείς ποσότητες. Θέλουμε λοιπόν να αφήσουμε και την πόρτα ανοιχτή για να βοηθήσουμε τρίτες χώρες που δυσκολεύονται να ε, διαχειριστούν ε, τα απόβλητα υδρουργύρου τους. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ καλό ε, επιχείρημα για την επιλογή της συγκεκριμένου οδού. Στην πρόταση αναφερόμαστε στις εισαγωγές υδραγύρου, ευθυγραμμίζονται με την σύμβαση της Μιναμάτα και εφαρμόζουμε κατάλληλο εργαλείο για τον περιορισμό των εισαγωγών υδραργύρου. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να απάντησα στις περισσότερες παρατηρήσεις. Θα κλείσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον εισηγητή για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φλόρεντς που μου απίφθενε την φιλοφρόνηση ότι είμαι τόσο νέος που δεν μπορώ να κρίνω. Αγαπητέ Φλόρεντς, μάλλον έχω περισσότερα χρόνια στην πλάτη μου από όσα ε, φαίνεται να υποθέτεις. Αλλά αυτό οφείλεται στην ε, διατροφή μου που είναι απολύτως χορτοφαγική. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα. Είχα την ευκαιρία να εξετάσω τις κόκκινες γραμμές και τα λοιπά των, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια για να λάβω υπόψη τις επικοδομητικές παρατηρήσεις των συναδέλφων μου, διότι είμαι πεπισμένος ότι για όλες και όλους μας η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος είναι θέμα προτεραιότητας. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι προσπάθειες για την μείωση όλων των κινδύνων που έρχονται από τον υδράγυρο είναι λίγο πολύ ανεπαρκείς και χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικά μέτρα και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Για να τα επιδείχουμε τα μέτρα αυτά πρέπει να διευρύνουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες κοινωνικο, ώστε κοινωνικο, κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις να μελετηθούν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, να δείξουμε το θάρρος, να εγκαταλείψουμε τη ζώνη μέσα στην οποία αισθανόμαστε άνετα και τις προκλήσεις να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες. Η δε στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παρακολουθείτε απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η οικονομική πολιτική της Ένωσης έχει οδηγήσει σε καινοτόμες λύσεις. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα παλαιά συνθήματα, ότι δήθεν η προστασία του περιβάλλοντος αντιβαίνει στις ανάγκες της ε, ε, βιομηχανίας και της οικονομίας. Ας αντιληφθούμε την περιβαλλοντική πολιτική ως πολιτική βιωσιμότητας, αηφορίας και βεβαίως η προστασία του μέλλοντος. Μέσα σε αυτά εντάσσεται και η προσπάθεια στήριξης των καινοτόμων ε, λύσεων της ε, ε, βιομηχανίας. Ένας κόσμος ο οποίος να είναι ασφαλής και για τα παιδιά μας και για τις μέλουσες γενιές. Αν λοιπόν είμαστε πραγματικά σοβαροί σε ό,τι αφορά την μείωση των εκπομπών υδραργύρου, πρέπει να θέλουμε ταυτόχρονα έναν κόσμο με λιγότερο υδράργυρο. Να κάνουμε λοιπόν φιλόδοξα βήματα, γιατί αλλιώς θα χαθούμε σε μια προσπάθεια κάποιων επιφανειακών διορθώσεων. Οι οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Καθήκον της περιβαλλοντικής πολιτικής οφείλει να είναι να δοθεί φωνή στις ε, ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και να μην επηρεάζεται από τις δυνατές φωνές των οικονομικών συμφερόντων. Μια προοδευτική κοινωνία θα πρέπει ωστόσο να είναι και μια, και μια λογική πρόκληση και για την βιομηχανία, για να γίνουν επενδύσεις σε καινοτομία, διότι το περιβάλλον και η οικονομική πρόοδος συμβαδίζουν. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε στο 12 παρα 5. Έναν πλανήτη έχουμε στη διάθεσή μας και οφείλουμε να τον προστατεύσουμε με συνέπεια. Ευχαριστώ για την ε, επικοδομητική σας στάση, αναμένω τη συνεργασία μαζί σας και σε, σας εύχομαι σε όλους και όλους καλές θερινές διακοπές, να μπορέσετε να ξεκουραστείτε για να επανέλθουμε στην εργασία μας το φθινόπωρο και να μπορέσουμε και να επισκευάσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Θα δώσω το λόγο πάλι στην κυρία Ουίνινγκ όπως ζήτησε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυσμόνησα να ευχαριστήσω βεβαίως τον εισηγητή μέσα στην ε, έντονη προσπάθειά μου να απαντήσω. Η συνεργασία του ήταν πολύ σημαντική και για την ε, ταχύτητα της πρόθεσης του θέματος ώστε να είμαστε έτοιμες για την κύρωση και της σύμβασης. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Σιγητά καθώς και τους κύριους Σιγητάς. Ο Προεδρεύων. Ευχαριστώ και συγχαίρω τον νεαρό εισηγητή κύριο Εκ. Πριν να προχωρήσω στο επόμενο ε, θέμα, σας υπενθυμίζω ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να έχουν κατατηθεί μέχρι τις 13 Εβδόμου στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 13 Δεκάτου και θα, θα έρθουμε τώρα στο επόμενο θέμα, όπως θύμισε και ο πρόεδρος μας Λαβία προηγουμένως, δεν θα συζητήσουμε με την Όλαφ την Υπηρεσία Καταπολέμησης Απατών, διότι θα είδατε την προηγούμενη εβδομάδα την Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Philip Morris International που δεν ανανεώθηκε η συμφωνία αυτή δεν θα έχει λοιπόν νόημα να γίνει η συζήτηση που είχε προβλεφθεί για το σημερινό απόγευμα. Θα έρθω λοιπόν στο 22 ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ενρικ Βέγγενερ που είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Σε Επιτροπή Θα ήθελα λοιπόν να ε, ευχαριστήσω πρώτα την Επιτροπή σας που μας προσεκάλεσε, που με προσκάλεσε μάλλον να κάνω, με συγχωρείτε διακόπτη ο Προεδρεύων, όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα να το πράξουν ησύχως για να μπορέσουμε να απολαύσουμε κάποια ησυχία καθώς θα μιλεί ο προσκεκλημένος μας. Σας ευχαριστώ. Ορίστε κύριε. Ευχαριστώ την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την πρόσκληση να παρουσιάσω το νέο μηχανισμό επιστημονικών συμβουλών. Λέγομαι Ρέγνερ και είμαι επικεφαλής της ε, Ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου επιστημονικών συμβουλών. Είμαι καθηγητή για ζωονόσους και ασφάλεια τροφίμων. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρο τη επαγγελματική μου σταδιοδρομία μελετώντα τα επιστημονικά τις επιστημονικές ενδείξεις για την Επιτροπή σας αλλά και για άλλες σημαντικές νομοθετικά επιτροπές όπως για προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια τροφίμων. Είμαι και αντιπρόεδρος του Πολυτεχνείου στην Δανία. Όμως, βρίσκομαι ενώπιον σας σήμερα, ιδίω με την ιδιότητά μου του νεοδιοριστέντος Προέδρου του High Level Group για Scientific Advice και έχω και μαζί μου και τρία μέλη της γραμματείας της Επιτροπής αυτής, Καρβάλιο, που σίγουρα μην γνωρίζετε, Μιμπρέη και Γιάν Μάρκο Μιούλερ. Ελπίζω λοιπόν με την παρουσίαση που θα σας κάνουμε να μπορέσω να δείξω στην Επιτροπή σας για ποιο λόγο θεωρώ ότι ο μηχανισμός επιστημονικών συμβουλών είναι μια σημαντική προσθήκη στους οργανισμούς που προσφέρουν επιστημονικές συμβουλές στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να αλλάξει η διαφάνεια πατών το κουμπί, αλλά δεν ανταποκρίνεται. να λέω τότε επόμενη διαφάνεια και να το κάνετε εσείς. Ah, you also have to turn it. Α, πρέπει βεβαίω να το βάλω μπροστά το μηχάνημα. Ευχαριστώ για την τεχνική σας υποστήριξη. Ο μηχανισμός λοιπόν βασίζεται σε μια μακρά ιστορία χρήσης των επιστημονικών δεδομένων για την λήψη αποφάσεων πολιτικής, ξεκινώντας από την ε, ίδρυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών και του συστήματος υποστήριξης των ευρωπαϊκών θεσμών και με τα προγράμματα πλαίσια τα οποία έχουν ε, αναπτύξει πολλές από τις ε, επιστημονικές μελέτες που έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε πολλούς τομείς πολιτικής. Υπάρχει και ένας αριθμός αποκεντρωμένων οργανισμών ήδη από τη δεκαετία του 90 και επίσης η Επιτροπή ΣΤΟΑ που ε, ιδρύθηκε για να υποστηρίζει την εργασία του Κοινοβουλίου το 2012 δημιουργήθηκε ο μηχανισμός και Αυτόν, αυτός είναι ο ρόλος του μηχανισμού, δηλαδή η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων. Αποφασίστηκε από τον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ ότι πρέπει αυτό να μας προβληματίσει και να αναπτύξουμε εκ νέου την λειτουργία αυτή μέσα σε ένα νέο μορφότυπο. Γι' αυτό ο Επίτροπος Μοέντας εκλήθη να προτείνει νέο μηχανισμό που να αναλάβει τα καθήκοντα αυτά παροχής επιστημονικών συμβουλών σε υψηλό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λειτουργήσει επίσης σαν συντονιστικό όργανο των επιστημονικών συμβουλών σε όλους τους τομείς των ε, ε, ευρωπαϊκών αποφάσεων. Τα αποτελέσματα του προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν τελικώς η θέσπιση του μηχανισμού παροχής επιστημονικών συμβουλών, το βλέπετε αυτό στο κέντρο της διαφάνειας, αποτελείται από υψηλή ομάδα, από υψηλού, υψηλού επίπεδου μάλλον ομάδα εργασίας επιστημονικών συμβούλων και μια γραμματεία που παρέχει την επιχειρησιακή υποστήριξη στην High Level Group. Συγκρίνεται λοιπόν με τον προηγούμενο ρόλο που έπαιζε ο Επιστημονικός Σύμβουλος με ευρύτερες αρμοδιότητες και ευρύτερο δυναμικό για να μπορεί να αντιμετωπίζει πιο περίπλοκα ζητήματα και βέβαια και περισσότερο όγκο εργασίας. Ο μηχανισμός ανταποκρίνεται σε αιτήματα που του υποβάλλονται από τον Πρόεδρο και το Σώμα των Κοσμητόρων Αυτά όλα πηγαίνουν μέσω του Επιτρόπου ΜΟΕΝΤΑΣ και αναφέρεται στον Πρόεδρο και στο Σώμα των Κοσμητώρων πάλι μέσω του Επιτρόπου ε, Μοέντας. Προσφέρει δεδομένα από συνεργασία με επιστημονικές οργανώσεις από τη, που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και από την επιστημονική κοινότητα. Στην βάση της ιδέας ότι θα πρέπει να μπορούμε να βασιζόμαστε σε όλα τα επιστημονικά δεδομένα που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας, πέραν των παραδοσιακών ορίων της επιστήμης και μέσα σε μια ολιστική επιστημονική αντιμετώπιση για κάθε θέμα το οποίο μας απασχολεί στις δραστηριότητές μας. Στην διαφάνεια αυτή βλέπετε φωτογραφία των μελών της ε, High Level Group επιστημονικών συμβούλων. Βλέπετε ε, ε, έξω αριστερά τον κύριο Σέντρικ Βιδιανή, ο οποίος είναι γνωστός Γάλλος μαθηματικός, η κυρία Φορτουνάτο, που είναι και αντιπρόεδρος, Πορτογαλίδα επιστήμων, πολύ γνωστή στην πατρίδα της, ο Ρόλφ Ντίτερ Χόερ, μέχρι πρόσφατα ήταν προ, ε, διευθυντής του ΣΕΡΝ, πυρηνικός φυσικός. Γιάννος Πουσνίκη, Πολωνός, ε, της Μοριακής Βιολογίας. Η Τζούλια Σλίνγκο είναι Βρετανίδα μετεωρολόγος, επικεφαλής της ε, μετεωρολογικής υπηρεσίας και εγώ ο ίδιος που είμαι ο πρόεδρος που ασχολούμαι όπως εξήγησα με την ασφάλεια τροφίμων. Αυτά τα πρόσωπα αποτελούν την ομάδα. Όπως θα δείτε καλύπτουμε πολλούς τομείς επιστημονικής δραστηριότητας και η φιλοδοξία μας είναι να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με θέματα και ερωτήματα σε κάθε τομέα πολιτικής, να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα επιστημονικής ε, συνεισφοράς. Τα καθήκοντα του μηχανισμού παροχής επιστημονικών συμβουλών και της High Level Group είναι να απαντούμε, να προσφέρουμε δηλαδή επιστημονικές συμβουλές για την ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθετική διαδικασία ανα πάσα στιγμή και σε κάθε τομέα πολιτικής. Μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο το καθήκον αυτό και όπου υπάρχει ανάγκη άμεση χορήγηση επιστημονικών συμβουλών. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να επικαλυπτόμεθα με υφιστάμενες επιστημονικές συμβουλές που προέρχονται από τον μεγάλο αριθμό επιτροπών, επιτροπών εμπειρογνωμόνων. Θα πρέπει λοιπόν πάντοτε η δική μας εργασία να είναι συμπληρωματική. Να μην επαναλαμβάνει δηλαδή πράγματα τα οποία ήδη είναι διαθέσιμα. Και όπως πρέπει σε κάθε επιστημονική αξιολόγηση θα πρέπει πάντοτε να θεμελιώνουμε και τις επιστημονικές συμβουλές που παρέχουμε. Επίσης μας ζητείτε να είμαστε προδραστικοί, δηλαδή να εντοπίζουμε ε, τομείς όπου θα χρειαστούν επιστημονικές συμβουλές να ε, κάνουμε συστάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων και αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να ενισχύουμε συνέργειες με άλλες δομές παροχής επιστημονικών συμβουλών. Θα ήθελα να τονίσω επίσης περισσότερο λίγο αυτό το τελευταίο που είπα, διότι θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει έναν από τους τομείς όπου έχουμε το δυναμικό να επιφέρουμε τις πλέον σημαντικές αλλαγές στην ε, δυνατότητα, στην ικανότητα μάλλον, στην ευρωπαϊκή ικανότητα παροχής επιστημονικών συμβουλών για αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν τις ε, πολιτικές αποφάσεις. Είμαστε και σε επαφή με όλες τις ε, οργανώσεις πανεπιστημιακών για να συνεργαστούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη της δυνατότητας χωρίς επιστημονικών συμβουλών για τις λήψεις αποφάσεων. Μέχρι τώρα ο τομέας ήταν κατακαιρματισμένος σε πολλές χώρες μέλη και στην δική μου οι πανεπιστημιακές οργανώσεις και ενώσεις οι πανεπιστημιακές ενώσεις γενικότερα, δεν έπαιζαν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση, παροχή πληροφοριών για, τις, για τη διευκόλυνση των πολιτικών ε, συζητήσεων και αποφάσεων στην βάση των βέλτιστων επιστημονικών γνώσεων. Τώρα, με την θέσπιση του μηχανισμού του ΣΑΜ, και συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Πανεπιστημιακές Ενώσεις ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διαρθρώσουμε με τέτοιο τρόπο ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη ώστε να παίξει ενεργότερο ρόλο στην παροχή επιστημονικών δεδομένων και συμβουλών για τους makers από όλες τις πηγές που θεωρούνται ανεξάρτητες αλλά και δραστηριοποιούμενοι στα υψηλότερα επίπεδα της επιστημονικής γνώσης. Εκτός του ότι είμαστε ανεξάρτητοι, πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό του χαρακτήρα του μηχανισμού μας, είμαστε και διαφανείς. Κάθε τι που κάνουμε θα γίνεται κοινό κτήμα, έχουμε ιδρύσει και ιστοσελίδα για να βοηθεί ακριβώς να ενισχύει τις προσπάθειες διαφάνειας. Τα πρακτικά των συνεδριάσεών μας και όλα τα σχετικά έγγραφα που περιγράφουν το έργο το οποίο κάνουμε και σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει το κάθε θέμα, αλλά και τα συμπεράσματα για κάθε θέμα, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε να μπορεί να τα ε, διερευνά κάθε ενδιαφερόμενος. Ποια θέματα μας έχουν απασχολήσει. Αρχικώς εγκύψαμε σε δύο θέματα για επιστημονική αξιολόγηση. Το ένα είναι η κυβερνοασφάλεια, όπου δεν θα επεκταθώ πολύ, στην δική σας εδώ επιτροπή. Το άλλο θέμα, ίσως να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για σας και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να επεκταθώ λίγο περισσότερο και να εξηγήσω τι έχουμε κάνει και να σας κάνω και μια εισαγωγή στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Το θέμα λοιπόν αυτό για το οποίο μιλώ τώρα είναι το κλείσιμο του κενού μεταξύ των πραγματικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος από ελαφρά οχήματα και των δοκιμασιών σε εργαστήρια. Το καθήκον αυτό μας ζητήθηκε να το αναλάβουμε από τον Επίτροπο Κανιέτε, μετά από αίτηση μάλλον του κ. Κανιέτε στον Επίτροπο Μοέντας και βασισμένη στην αίτηση αυτή συντάξαμε ένα scoping paper το οποίο οριοθετούσε στην βάση το είδος εργασίας που θέλαμε και μπορούσαμε να αναλάβουμε σε διάλογο με τον Επίτροπο καταλήξαμε ότι το έργο αυτό θα πρέπει όντως να επιτελεστεί. Το scoping paper οριοθέτησε το πεδίο εφαρμογή του έργου μας με δύο παράλληλες κινήσεις από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφενό να διασφαλίσουμε ότι τα νέα προγράμματα δοκιμασιών για εκπομπές καυσαερίων θα είναι όσο γίνεται αντιπροσωπευτικότερο του πραγματικού κόσμου για τις εκπομπές διοξιδίου του ανθρώπου και από την άλλη μεριά να εξετάσουμε την χρήση ευρείας κλίμακος δεδομένων κατανάλωσης καυσίμων για να καταλήξουμε σε κάποιες εκτιμήσεις που να είναι όσο γίνεται πλησιέστερες στον πραγματικό κόσμο. Τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν τον ΣΑΜ εν προκειμένου είναι ποια είναι η επιστημονική βάση για την βελτίωση της μέτρησης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος ελαφρών οχημάτων και κατανάλωση καυσίμων για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αξίες που να αποδίδουν τον πραγματικό κόσμο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιες ε, προσεγγίσεις μπορούν να εκτιμηθούν και σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την διαφάνεια και ποιες πρόσθετες εργασίες επιστημονικές και αναλυτικές θα χρειαστούν. Άρα θα υποβάλουμε μία στέρεα θεμελιωμένη επιστημονική προσέγγιση στα επόμενα χρόνια. Για να χρησιμοποιηθεί μάλλον στη λήψη αποφάσεων τα επόμενα χρόνια. Το χρονοδιάγραμμα της εργασίας μας προβλέπεται το εξή. Για το θέμα αυτό. Το βλέπετε άλλωστε στη διαφάνεια. Όταν δεχθήκαμε το scoping paper τον Φεβρουάριο αποφάσισαμε ότι θα καταθέσουμε γνωμοδότηση τον Οκτώβριο. Άρα επαρκές χρονικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί η ακρίβεια της διαδικασίας διεξαγάγαμε και εξακολουθούμε να διεξάγουμε έρευνες και συλλογή δεδομένων μεταξύ αυτών και με επίσκεψη σε μια από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Ίσπρα της Ιταλίας τον Ιούνιο Διεξήθη εργαστήριο με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί επιλέχθηκαν μετά από προσεκτική αξιολόγηση όλων των εμπειρογνωμόνων που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσώπων που έχουν αποδεδειγμένα μεγάλη επιστημονική αξία και το έργο τους είναι συμπληρωματικό, άρα θα καλύψει όλα τα σχετικά θέματα. Προσκλήθηκαν οι εμπειρογνώμονες στη Λισαβόνα να συμμετάσχουν σε εργαστήριο και έχουμε συλλέξει μεγάλο όγκο επιστημονικών δεδομένων από το δεύτερο αυτό. Τον Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών όπου θα προσκαλέσουμε τους stakeholder και εκτός της επιστημονικής κοινότητας για να μας παράσχουν πληροφορίες για την ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου πριν να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο της γνωμοδότησής μας τον Οκτώβριο. Να λοιπόν με λίγες γραμμές ο τρόπος εργασίας μας. Συλλογή της διαθέσιμης βιβλιογραφίας όπως γίνεται όταν κάνει κανείς επιστημονικές αξιολογήσεις, εργαστήρια εμπειρογνωμόνων, επιλεγμένων εμπειρογνωμόνων, ε, στην βάση της επιστημονικής τους αξίας. Αυτές οι επιστημονικές συγκεντρώσεις, συναθρήσεις ήταν πολύ χρήσιμες για μας. Μετά διάλογος με τους ενδιαφερομένους φορείς και τέλος σύνταξη και έγκριση του κειμένου γνωμοδοτήσεω. Με το παράδειγμα αυτό ελπίζω να μπόρεσα να σας δείξω με ποιον τρόπο προτιθέμεθα να εργαστούμε για τα θέματα αυτά που είναι μια σημαντική περιπλοκότητα και απαιτούν μια πολυτομιακή ε, επιστημονική προσέγγιση. Σκεπτόμενος τα ενδιαφέροντα της Επιτροπής σας, θα σας παραπέμψω και στην ιστοσελίδα μας όπου θα δείτε ότι έχουμε εργαστεί και σε ένα τρίτο θέμα σε πολύ συντομότερο χρονικό πλαίσιο όχι για να συντάξουμε γνωμοδότηση αλλά μάλλον για να δώσουμε μια εξήγηση επεξηγηματικό σημείωμα για το θέμα της γλυφοσάτης για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο και τον Αρμόδιο Επίτροπο για την κατάσταση στην οποία, για την πρόοδο στην οποία βρίσκονται οι σχετικές επιστημονικές μελέτες. Με τα λόγια αυτά ολοκληρώνω την παρουσίασή μου και πολύ ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κανείς συνάδελφος το λόγο. Όχι. Δεν ζητά κανείς το λόγο. Ρωτήσεις, τίποτα. I'm going. Η κυρία Γκέρλινγκ. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω για τη σχέση ή αν υπάρχει σχέση με το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει για την ώρα, αλλά πώς θα μπορούσε να υπάρξει εάν εξετάσετε ας πούμε θέματα τα οποία και εμείς εξετάζουμε και πώς και αν θα μπορούσατε να μας δίνετε και εμάς σε πληροφορίες. Βλέπετε ε, δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει, έχετε και αυτό το ρόλο το συμβουλευτικό προς το Κοινοβούλιο. Merci beaucoup. Ναι, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ έλεγα πως όχι άμεσα, αλλά προφανώς οι γνωμοδοτήσεις και μελέτες που προέρχονται από τον Μηχανισμό Επιστημονικής Συμβουλής θα είναι διαθέσιμες ώστε να ε, ε, χρησιμοποιηθούν στις συζητήσεις και στις αποφάσεις που λαμβάνει το Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε την πολιτική συζήτηση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται λοιπόν εντό Κοινοβουλίου. Έχουμε ανταλλαγές απόψεων με την Επιτροπή ΣΤΟΑ. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε τις πολιτικές συζητήσεις που γίνονται για τους τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε κι εμείς ώστε οι συμβολές μας να είναι όσο γίνεται πιο βοηθητικές και επικοδομητικές για στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Merci. Σας ευχαριστώ. Εάν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, κυρία Γκροστέτ, παρακαλώ. Ναι. Εξαρτάστε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε προσωπικά να ζητήσουμε μια επιστημονική γνωμοδότηση. Ας πούμε, δουλεύουμε για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ένα εξαιρετικά λεπτό και συναισθηματικό θέμα που όμως εμείς θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο γίνεται πιο βάσιμη, διαλογημένη και αιτιολογημένη θέση. Ας πούμε, για ένα τέτοιο θέμα θα μπορούσατε να μας δώσετε μια γνωμοδότηση που να μπορούσε να μας διαφωτίσει πόσο προηγείται και για ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ναι, σας ευχαριστώ. Κατά την αντίληψή μου, είτε θα πρέπει να απαντήσουμε σε αιτήματα της Επιτροπής, είτε αυτενεργούμε. Και όταν αυτενεργούμε έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε θέματα όπου μπορούμε, ε, ε, κατά τη γνώμη μας, να προσθέσουμε σημαντική επιστημονική γνώση. Στο πλαίσιο των ενδοκρινικών διαταρακτών γνωρίζω ότι ήδη γίνεται πολλή δουλειά Προσωπικώς δεν γνωρίζω κατά πόσον εμείς μπορούμε να προσθέσουμε κάτι. Πάντως, μαζί με πολλά άλλα θέματα που συζητώνται εξετάζονται, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και αυτό. Σίγουρα είναι από τα θέματα που μας απασχολούν και τα προσέχουμε. Σίγουρα μπορούμε και σε διάλογο με τη ε, διάφορες, ε, τα διάφορα ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, θα μπορούσαμε να τους καλέσουμε να ασχοληθούν με κάποιο θέμα. Γιατί αν, ε, ας πούμε, όπως είπα και στην εισήγησή μου, μπορεί εμείς να αναλάβουμε 5, 6 και μέχρι 6, ας πούμε, θέματα ετησίως. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα δύσκολα ζητήματα για τα οποία απαιτείται περαιτέρω εργασία για να μπορέσουμε να κάνουμε επιστημονικές αξιολογήσεις η δύναμή μας λοιπόν είναι ότι αν καταφέρουμε να έχουμε αυτόν τον επικοδομητικό και δομημένο ε, διάλογο με όλα τα επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο στέρεες βάσεις για να συμβάλλουμε στην ενημέρωση την επιστημονική σας. Σίγουρα λοιπόν και τα ερευνητικά ιδρύματα μπορούν να συμβάλλουν στην ενημέρωση πριν τη λήψη αποφάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Όχι. Ωραία, λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για αυτήν την παρουσίαση που μα κάνατε. Και τώρα θα περάσω στο επόμενο σημείο, το υπερθόν 23 όπου έχουμε να κάνουμε με ένα ψήφισμα που έχει κατατεθεί για τα τρανς Οι συνεισηγητές δεν είναι εδώ, αλλά είναι η κυρία Σόμερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι θα μου δώσετε τόσο γρήγορα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κρίμα που συζητάμε το θέμα αυτό σήμερα που τόσοι συνάδελφοι ε, έχουν να κάνουν κάτι άλλο. Αλλά χαίρομαι που μπορέσαμε να συμφωνήσουμε πάνω στο, στην πρόταση ψηφίσματος αυτήν. που έχει να κάνει με τα τρανς λιπαρά στα τρόφιμα. Χαίρομαι που η Κομισιόν ε, υπέβαλε την πρόταση την οποία περιμέναμε νωρίτερα, το Δεκέμβριο του 2015 στην έκθεσή της η Κομισιόν δείχνει τη σχέση ανάμεσα σε καρδιακιακές νόσους και την ε, αυξημένη πρόσληψη τρανσλιπαρών οξέων. Και σας ευχαριστώ για την ε, έκθεση, διότι στην ε, συζήτηση σχετικά με την οδηγία για τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, για την ενημέρωση των κατανοτών, δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά τα τρανθλιπαρά οξέα στα τρόφιμα, διότι δεν είχαμε αρκετές γνώσεις τότε, δεν γνωρίζαμε. Έχει νόημα ο καταναλωτής ξέρει τι είναι τα τρανσλιπαρά Είναι δυνατόν να έχουμε σχετική επισήμανση στα τρόφιμα ε, ή να ορίσουμε ανώτατες τιμές επιτρεπόμενης πρόσληψης. Έτσι λοιπόν αναθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ε, έκθεση Ε, υπήρχαν όμως επιθυμίες ε, για περιορισμό της ε, πρόσληψης τρανσλιπανών στα τρόφιμα. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στις καρδιακικές παθήσεις και την κατανάλωση τρανσλιπανών Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε σημαντική μείωση των καρδιακών παθήσεων και βλέπουμε ότι το πρόβλημα κυρίως ε, σχετίζεται με συγκεκριμένα τρόφιμα. Η Κομισιόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια ανώτατη τιμή για ε, τα τρανστιπαραοξέα είναι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή και δεν είμαι η μόνη. Αρκετοί συνάδελφοι συμφωνούν με μια τέτοια προσέγγιση για τον λόγο ότι το πολύ το 1 τρίτο των πολιτών μας ε, γνωρίζει τι είναι τα τρανσλιπαρά οξέα. Γι' αυτό η σχετική επισήμανση στα τρόφιμα δεν θα είχε νόημα. Διότι ε, οι περισσότεροι δεν ε, αναγνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές, οπότε ήταν πιο χρήσιμο να υπάρχει ανώτατη τιμή περιεκτικότητα στα τρόφιμα. Εκτός από την Επιτροπή ε, θα λάβει και το Συμβούλιο ε, προφορική ερώτηση από εμά ε, και αναρωτιέμαι αν συμμερίζεται τη θέση μας. Πρέπει όμως να δώσουμε και αρκετό χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσει τις επιπτώσεις ανώτατων τιμών στον βιομηχανικό τομέα στους παραγωγούς και μάλιστα στα διάφορα μεγέθη ε, επιχειρήσεων. Και επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα του μέτρου αυτού. Ε, δεν είναι πολύ απλό, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που θεωρούν ότι δεν χρειαζόμαστε νέα μελέτη αντικτύπου και ότι θα πρέπει αμέσως να εφαρμόσουμε ε, τις ε, τιμές αυτές. Εγώ θα ήθελα όμως να υποβάλω τροπολογία που να ζητάει νέα μελέτη αντικτύπου. το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε με τα οξέα που δημιουργούνται κατά την ε, παρασκευή τροφίμων. Για παράδειγμα, όταν φτιάχνω τηγανιτές πατάτες, ε, με τη διαδικασία ε, του τηγανίσματος παράγονται οξέα. Πώς θα χειριστούμε λοιπόν αυτά. Θα έχουμε και εδώ κάποια ανώτατη τιμή τα μη συσκευασμένα ε, φρέσκα νοπά τρόφιμα ε, θα πρέπει να περιέχουν ε, επισήμανση και εάν ορίσουμε οριακές τιμές και για τέτοιες ομάδες προϊόντων, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον τομέα που παρασκευάζει φρέσκα τρόφιμα. Κάτι τέτοιο μπορεί να φαίνεται από τα συστατικά του προϊόντος, ε, αλλά ε, θα πρέπει να αναφέρεται και η διαδικασία παρασκευής των τροφίμων. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε νέα μελέτη αντικτύπου. Επίσης, ε, δεν βρίσκω πολύ σκόπιμο να συνδέουμε τα τρανσλιπαρά οξέα με όλες τις ασθένειες του κόσμου, όπως γίνεται στο σχέδιο ψηφίσματος. Ε, λίγες ε, είναι οι ασθένειες παθήσεις ε, που, όπου έχει τεκμηριωθεί η σχέση με την κατανάλωση τρανσλιπαρών οξέων, με την ενδομετρίωση. Από ό,τι γνωρίζω δεν, δεν συνδέει καμία μελέτη την κατανάλωση τρανσλιπαρών Επίσης, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα τρανσιπαρά οξέα που υπάρχουν ε, ε, από τη φύση, όπως ε, στο γάλα ή στο κρέας. Εδώ θα πρέπει να τα παραβλέψουμε. Εδώ υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των συνεισηγητών. Μερικοί πιστεύουν ότι αυτά τα Φυσικά, τρανς, λιπαρά, οξέα δεν θα πρέπει να τα αναφέρουμε, διότι δεν μπορούμε εδώ να θέσουμε ε, τιμές, ε, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνουν πολύ κρέας και έτσι αυξάνουν την ε, πρόσληψη τρανς, λιπαρών, οξέων. Τα φυσικά τρανς λίπαρα οξέα, άλλωστε είναι όμοια με αυτά που ε, προστίθονται στα τρόφιμα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να καθορίσουμε ποια είναι τα οξέα και σε ποια τρόφιμα περιέχονται. Και μια τελευταία παρατήρηση. Δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε ότι με την ε, εισαγωγή μιας ε, ανώτατης τιμής θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλα λιπαρά οξέα, τα οποία μπορεί να μην είναι πολύ υγιεινά, θα πρέπει να αναφέρονται στην συσκευασία, αλλά μπορεί τελικά να ε, αντικαταστήσουμε το ένα βλαβερό ε, συστατικό με ένα άλλο. Ε, και θα πρέπει βέβαια να έχουμε υπόψη μας τη συζήτηση περί βιωσιμότητας, η οποία θα πρέπει να μας απασχολήσει διότι η εναλλακτική λύση για τα οξέα είναι το φινικέλαιο και Γνωρίζουμε ότι ε, η αντικατάσταση τρανσλιπαρών οξέων από ε, φινικέλαιο μπορεί να οδηγήσει σε ε, έλλειψη αυτού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σόμερ. Ευχαριστώ. Και τώρα... Σας ευχαριστώ πολύ. Παίρνω το λόγο ε, εκ μέρους της κυρία Αρπού που είναι συνεισηγήτρια ε, και το κάνω αυτό. Ευχαρίστω διότι συμφωνώ σε πολλά μαζί της. Η κυρία Σόμερ ε, ήδη ανέφερε πολλά θέματα με τα οποία συμφωνούμε και εμείς. Τα τρανσλιπαραοξέα αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Στο ψήφισμα αυτό ζητάμε την θέσπιση ανώτατων τιμών για τα βιομηχανικά τρανσλιπαραοξέα στα τρόφιμα. Ήδη υπάρχουν ε, ε, λέτες σχετικά με ε, τις τιμές πρόσληψης και βλέπουμε ότι ο περιορισμός της κατανάλωσής τους μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό καρδιακτικών νοσημάτων. Και μάλιστα τα αποτελέσματα αυτά είναι ορατά ήδη μέσα σε λίγα χρόνια. Έχουμε επικεντρωθεί στα βιομηχανικά τρανς και όχι αυτά που, εμφανίζονται φυσικά, που εμφανίζονται στη φύση τα τρόφιμα με ε, τα υψηλότερα ποσοστά τρανς λιπαρών οξέων, ε, είναι τα μπισκότα, τσίπς, ε, διάφορα τέτοια σνακ τα οποία καταναλώνονται από πολύ κόσμο και λόγω της χαμηλής τιμής τους. Ο περιορισμός των βιομηχανικών τρανς λιπαρών οξέων Ε, θα πρέπει να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις ακριβώ ε, στην κατηγορία του πληθυσμού ε, που έχει κακές συνήθειε ως προς την διατροφή. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ περιορισμένη η γνώση των πολιτών σχετικά με τις επιπτώσεις των τρανσιπανών στην υγεία και θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα patchwork νομοθεσιών. Λείπουν λοιπόν εναρμονισμένες διατάξεις και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόληψη καρδιακών παθήσεων. Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει τα συμπεράσματα της δικής της έκθεσης, να ορίσει δεσμευτικά όρια για τα τρανσλιπαρά οξέα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε και την ε, συμφωνία ΣΥΤΑ μετά την ε, TTIP ε, και χρήσιμο θα ήταν να δούμε τι κάνει η Αμερική και αν μπορούμε να εφαρμόσουμε τη λύση που έχουν επιλέξει εκεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο θα έχει η κυρία Φεντερίκ Ρίξε, ξανόματος της Άλντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο ψηφίσματος που έχουμε επιτάπητο σήμερα κατατέθηκε από τις 8 πολιτικές ομάδες, όλες δηλαδή, Πρόκειται για μια κοινή διαπίστωση και κοινή βούληση από πλευρά τη Επιτροπή μα και ελπίζω και του Κοινοβουλίου να μειωθεί η κατανάλωση των ε, τρανσλιπαρών οξέων. Γιατί ε, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση. Είναι η προτεραιότητα του Κοινοβουλίου μα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το λέμε νομίζω και στην πρώτη, πρώτη παράγραφο ότι τα λιπαρά οξέα συνδέεται με μια ολόκληρη σειρά ασθενειών. Ε, συμφωνώ με την κυρία Σόμερ ότι ίσω θα πρέπει κάπω να τακτοποιήσουμε τα εκτιμώντα. Όλα αυτά βρίσκονται στο εκτιμώντα ΖΕ. Μιλάμε για τι καρδιακέ παθήσει, αυτό είναι προφανέ, για την ε, ε δεν υπάρχει παχυσαρκία όμως, <laughs> όλος παραδόξος, οπότε σίγουρα θα κάνουμε εδώ μια δροπολογία. Ήδη είχαμε κρούσει το κόδωνα του κινδύνου πριν από 10 χρόνια ως εισηγήτρια για την οσιρότητα αυτών των λιπαρών οξέων σε μια έκθεση για την παχυσαρκία. Εν τω μεταξύ και παρά όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει στις 17 Μαρτίου μάλιστα τελευταία φορά το συζητήσαμε για το πρόγραμμα δράση της Επιτροπής θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν αρκετά γρήγορα. Εξελίσσονται ναι, αλλά όχι αρκετά γρήγορα και, όχι συντονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που προχωρά όμως είναι αυτές οι διάφορες ασθένειες όπως η παχυσαρκία. Διάβαζα πριν μια πρόσφατη μελέτη που έλεγε Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των λιπαρών οξέων στους νέους εφήβους που μπορεί να καταναλώσουν μέχρι και καθημερινά 10 γραμμάρια λιπαρά οξέα μέσω της κατανάλωσης ε, junk food, ε, παλιο, ε, παλιοφαγητών δηλαδή, έτοιμων μπισκότων. 10 γραμμάρια είναι, είναι τρεις φορές περισσότερο από το ανώτατο κατόφλι και το είχα αναφέρει και στην τελευταία μας συζήτηση. Η Δανία είναι στο προμαχών για αυτό το, στην καταπολέμηση, αλλά και η Ουγγαρία, η Λετωνία και η Αυστρία. Πέρα από τα όσα δηλαδή μπορεί να αποφασίσουμε, εκστρατείες ενημέρωση είναι απαραίτητε και ιδιαίτερα για τους νέους που είναι ο, κατεξοχήν στόχος. Σημείωσα σήμερα το πρωί γιατί ακούσαμε τον ε, Σλοβάκο Υπουργό Υγείας τον προεδρεύοντα, τον Τόμας Ντρούκερ, που έκανε ένα άνοιγμα σε αυτή την καταπολέμηση της κατανάλωσης λιπαρών οξέων, να ενισχύσουμε τις εθνικές πρακτικές, είπε, σε θέματα αναδιατύπωσης των προϊόντων. Εθνικές πρακτικές, ναι, το είπα και εγώ, αλλά δεν αρκεί και είναι καλύτερο αν αυτές οι δράσεις γίνουν συντονισμένα και εναρμονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό λέμε και στην παράγραφο 6 νομίζω του ψηφίσματος. Εντάξει, δεν το επαληθεύσω στο ψήφισμα αυτό. Άλλο θετικό στοιχείο στο κείμενό μας είναι το γεγονός ότι αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα στις τρεις επιλογές, υποχρεωτική ετικετοθεσία, αξίες, οριακές αξίες, εθελοντικές συμφωνίες, όπως τα έχει πει και η Κομισιόν στην εκθεσή της του Δεκεμβρίου. Εγώ προσωπικά θα ήμουν υπέρ της θέσπισης μιας ε, οριακής τιμής για 100 γραμμάρια λιπαρής ε, ε, ουσίας, όπως εδώ στην παράγραφο 8 νομίζω, που λέμε πολύ συγκεκριμένα να υποχρεωτικά όρια σε σχέση με την ύπαρξη των λιπαρών οξέων. Συμμερίζουμε επίσης επικρίσεις όπως έχουν διατυπωθεί στην παράγραφο 7 τίποτα, δεν, δεν χρησιμεύει σε τίποτα να πνίγουμε τους καταναλωτές σε μια ροή τεχνικών πληροφοριών στην ετικέτα, όπου συχνά, όπως μας λένε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μπερδεύονται τελείως. Εγώ είμαι ολένα και πιο πεπισμένη ότι πρέπει να υπάρχει ένα απλοποιημένο σύστημα ε, σήμασης με χρώματα που θα πρέπει να γίνει με την συμμετοχή του κλάδου και το είπα και την περασμένη φορά όλα είναι και περισσότεροι στον τομέα των βιομηχανικών ε, δέχονται αυτήν τον αγώνα μεγάλη τομείς της ε, αγροτρο, αγροτοδιατροφικής ε, αλυσίδας για εξάλληψη με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτών των τρανσλιπαρών οξέων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Άρης για τη συμβολή σας και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπόιλαν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ξέρουμε ότι αυτά τα λιφπαρά είναι δολοφονικά. Υπάρχουν ένα σωρό αποδείξει που τα συνδέουν με μια μεγάλη σειρά ασθενειών ε, και είναι σε καθημερινά προϊόντα κατανάλωση. Είναι πολύ δύσκολο να τα αποφύγουμε. Μόνο στην Ολλανδία 10.000 κόσμος πεθαίνει από καρδιακέ παθήσεις ετησίω. Και βέβαια οι χαμηλότερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες είναι αυτές που καταναλώνουν τα trans είναι τα φθηνότερα και πιο κατεργασμένα τροφικά, διατροφικά προϊόντα. Επίση, δεδομένου του γεγονότο ότι βρισκόμαστε στην ασυνήθιστη θέση στην, ε, στην, ε, στην Ένωση, που είμαστε... Ε, πολύ συνδεμένοι με τη ΣΥΠΑ, αλλά εκεί είναι πολύ μπροστά Όσον αφορά το, το συγκεκριμένο τρόφιμα, ήδη έχουν διατάξει τους κατασκευαστές να τα αφαιρέσουν σε δύο χρόνια από όλα τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει κάποιες ευπρόσδεκτες υποδείξεις για μελλοντική δράση, αναγνωρίζει ότι πρέπει να τεθεί ένα νομικό όριο για βιομηχανικό και περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των καταναλωτή, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις ετικέτες. Δεν είναι σωστό, είναι, ε, ε, προκαλεί σύγχυση, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες και κυρίως επειδή οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι είναι αυτά τα λιπαρά οξέα. Θα ήταν, ε, εγώ δεν θα ήθελα να είναι στην ε, ετικέτα, γιατί ε, απλά δεν πρέπει να καταναλώνονται. Δεν πρέπει καν να είναι συστατικά των τροφίμων. Από το 2011 καλέσαμε την Κομισιόν να κάνει αυτή την έκθεση, αλλά να υποβάλει και νομοθετική πρόταση. Πιστεύω πως χρειαζόμαστε αυτή την ε, νομοθετική έκθεση. Χρειάζονται νομικά όρια για τα οξεία και πιστεύω πως ε, η μελέτη αντικτύπου είναι μια τακτική καθυστέρηση που έχουμε δει να χρησιμοποιείται και σε άλλους τομείς. Χρειάζεται λοιπόν μείωση στα λιπαρόξια. Ξέρουμε πως δεν είναι αδύνατον. Οι κατασκευαστές το κάνουν και μάλιστα εθελοντικά. Αυτό που χρειάζεται είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τη δημόσια υγεία και να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπόιλαν και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντονανό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να θυμίσω ότι στην έκθεση για τα λιπαρόξια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμιζε και σωστά τη σημασία των ε, τροφικών συνηθιών των νέων αλλά και των χαμηλών εισοδημάτων. Η ιδέα της ε, νέου κατάρτισης των καταναλωτών, όπως το έλεγε στο κείμενο, είναι με αυταπάτη. Το ψήφισμα αυτό εδώ οθεί την έγκριση ευρωπαϊκών ορίων όσον αφορά την παρουσία των λιπαρών οξέων αστείο τρόφιμα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για μέτρα αποτελεσματικό. Μάλλον, όμως να θυμίσουμε ότι επειδή η ευνοία αγορά εμποδίζει κάθε ποσοτικό ή ποιοτικό περιορισμό στην κυκλοφορία αυτών των τροφίμων, που είναι υποχρεωμένη να υιοθετεί η ίδια περιορισμούς στη θέση των κρατών. Η ιδια περιορισμού στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμιζε ότι σε περίπτωση υιοθέτηση εθνικών μέτρων από ένα κράτος, ο τομέας αυτός μπορεί να τιμωρεί το λόγω της εξωτερικής, του εξωτερικού ανταγωνισμού. Βλέπουμε σαφώς τα όρια της ενιαίας αγοράς. Εν πάση περιπτώσει, είναι θεμητό το να θέλουμε να μειώσουμε τους παράγοντες πρόκλησης καρδιακιακών παθήσεων, που είναι ένας από τους κύριους, τα κύρια αίτια θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. εγώ σας ευχαριστώ κυρία Αντωνανό και τώρα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν, στην κυρία Νικολακοπούλου. Yes, um, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν από τέσσερις περίπου μήνες η Κομισιόν ήρθε για να παρουσιάσει την έκθεση για τα τρανσλιπαρά οξέα. Θέλω να θυμίσω σύντομα τις κεντρικές πτυχές αυτής της έκθεσης που έδωσε πληροφορίες για την παρουσία λιπαρών οξέων στα τρόφιμα και γενικά στην δίαιτα των Ευρωπαίων περιέγραψε τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση λιπαρών οξέων και τους κινδύνους καρδιακών παθήσεων και συμπέρανε ότι το νομικό όριο για τα λιπαρά οξέα, τα βιομηχανικά παραγόμενα λιπαρά οξέα θα ήταν ένα, το πιο αποτελεσματικό μέτρο όσον αφορά τη δημόσια υγεία, την προστασία του καταναλωτή και τη συμβατότητα με την εσωτερική αγορά. Ωστόσο, η έκθεση αυτή σημείωνε στα απορίσματά της ότι θα έπρεπε να γίνουν περαιτέρω έρευνες και ανακοίνωνε την πρόθεση της Κομισιόν να διεξάγει εκτίμηση, εξολόγηση αντικτύπου συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας διαβούλευσης για το θέμα έτσι ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις στο εγγύς μέλλον. Η Κομισιόν ε, το Μάρτιο αλλά και σήμερα ε, ευχαριστημένη είναι που βλέπει ότι υπάρχει διακομματική στήριξη για ταχύες ενέργειες από πλευρά της Ένωσης ώστε να μειωθεί η πρόσληψη λιπαρών οξεών από τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Σας ε, διαβεβαιώνω ότι σήμερα λάβαμε υπόψη όλες τις ανησυχίες για αυτού του είδους τα λιπαρά οξέα και την ανάγκη για, τα, για γρήγορα αποτελέσματα. Σας διαβεβαιώνω ότι και Επίτροπος Αντριοκαΐτης ανησυχεί για αυτά τα λιπαρά οξέα ε, κατανοεί την ανάγκη για γρήγορη δράση. Ωστόσο, θα πρέπει να ξεχάσουμε την ε, δέσμευση αυτή τη Κομισιόν για την καλύτερη νομοθεσία, πράγμα που σημαίνει πολιτική ε, με βάση αποδείξει και μαρτυρίε. Ακόμα και αν υπάρχει ευρεία συνένεση για τα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε αποδείξει, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα δράσουμε με το πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο για να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η έκθεση για τα τραν λιπαρά εντοπίζει διάφορε πτυχέ που χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω ξέρω και ορισμένε από αυτέ αναφέρθηκαν μάλιστα και από κάποιου από του ευρωβουλευτέ στη συζήτηση του Μαρτίου αλλά και στη σημερινή συζήτηση, όπω για παράδειγμα πώς να εξασφαλίσουμε ότι μια πρωτοβουλία για τα τρανσλιπαρά δεν θα έχει δυσανάλογο αντίκτυπο το κόστος για τους ε, ε, ε, Παρασκευαστέ ε, τιμών ε, προϊόντων ε, και κυρίω για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, Αυτό το είπε η κυρία Σόμερ. Επίσης να δούμε ποιε αναλλακτικέ υπάρχουν για, να, για τα εν μέρη υδρογονωμένα έλαια που είναι ας πούμε, αυξημένη χρήση του του φινικελαίου μπορεί να έχει άλλες ε, αρνητικές επιδράσεις. Ε, ε, επίσης πρέπει όλες οι διατάξεις να μπορούν να επιβληθούν από καταλήλως από τις εθνικές αρχές ελέγχου. Ποιες ε, έχουμε αρκετές μεθοδολογίες ώστε να ορίσουμε το, την περιεκτικότητα σε τρανς λιπαρά, τρόφιμα, αλλά και να, να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα στα βιομηχανικά τρανς λιπαρά και τα ε, αυτοπαραγόμενα. να δούμε ε, ότι ε, θα δείτε μάλλον τις μελέτες μας ε, στις, πολύ σύντομα γιατί έχουμε κάνει τις σχετικές μελέτες και θα, δημοσιευθεί η, η μελέτη αντικτύπου για τα τρανσλιπαρά ε, σε λίγες εβδομάδες. Το έγγραφο αυτό προετοιμάστηκε από την DG Υγείας και τώρα συζητάτε με τις άλλες υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι μια συνοπτική αρχική εκδοχή ε, της, ε, του πλήρου, του πλήρους, της πλήρους μελέτης. Περιλαμβάνει περιγραφή του προβλήματος των μπλεκόμενων φορέων, εντοπισμό των στόχων που θέλουμε να επιτύχουμε, ανάλυση του πού θα πρέπει να ισχύσουν οι αρχές της, ε, και τηρούνται οι αρχές της ε, επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ανάλυση διαφόρων ε, πολιτικών επιλογών και επίσης ανάλυση των αντίστοιχων επιπτώσεων, καθώς και περιγραφή των αναγκών μας για στοιχεία, για πληροφόρηση και ποια είναι η στρατηγική που σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε. Θέλω να σας καταστήσω σαφές ότι αυτό εδώ δεν θα είναι επανάληψη της έκθεσης της Κομισιόν, αλλά θέλουμε να βασιστούμε στα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και στις αναλύσεις που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι ότι ε, έχουμε ήδη ένα χρονοδιάγραμμα ενδεικτικό. Ε, Μπορεί να γίνουν και άλλε συζητήσει εντωμεταξύ μέσα, στη, μέσα στην Κομισιόν. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη ε, αντικτύπου θα δημοσιευθεί στο χώρο, στον ιστοχώρο μας, ε, οπότε ενδιαφερόμενα μέρη θα δώσουν απόψει και κρατάει περίπου τέσσερι εβδομάδες. Εντωμεταξύ ε, σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε και ένα διαγωνισμό για την ε, μελέτη, ώστε να εμβαθυνθεί η ανάλυση μας για κάποιες πτυχές μια πρωτοβουλίας, ας πούμε αντίκτυπος της διάφορες πολιτικές επιλογές και αυτό θα διαρκέσει περίπου έξι μήνες. Τον επόμενο μήνα θα γίνουν και άλλες διαβουλεύσεις, ε, συμπεριλαμβανομένες μιας δημόσια διαβούλευση που θα κρατήσει 12 εβδομάδες. Αυτό μάλλον θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Επί τη βάση όλων αυτών των πληροφοριών, η μελέτη που θα ολοκληρωθεί και θα υποβληθεί στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο Ελέγχου στις αρχές του 2017. Και βεβαίως, ε, εάν επιβεβαιωθεί ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή δράση, τότε θα αναμένουμε ταχύες εξελίξεις. Φυσικά, ε, είναι πολύ σημαντική η ταχύτητα της δράσης, θα συνδέεται και με το είδος των νομικού ε, μέσου που θα επιλεγεί. Για παράδειγμα, θα ξέρετε πως αν ακολουθήσουμε την συνηθισμένη νομοθετική διαδικασία, αυτή κρατά περισσότερο από ότι ένα μέτρο μη νομοθετικό του τύπου της επιτροπολογίας. Αυτά επίσης θα τα εκτιμήσουμε προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη, όπως ε, τονίστηκε και από εσά ότι όσο γρήγορα, ενεργήσουμε τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα ωφέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά μπορώ να σας πω ενημερωτικά σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Νικόλα Κοπούλου κάποιες πληροφορίες για το ψήφισμα αυτό τώρα. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στις 12 και θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 29 Σεπτεμβρίου και κανονικά λοιπόν η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται για τη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο τα διάφορα. Δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε στα διάφορα. Απλά μια τελευταία πληροφορία ότι η επόμενη μας συνεδρίαση προβλέπεται για την 1η Σεπτεμβρίου από τις 9 στις 12.30. Επιτροπή Περιβάλλοντος εδώ λοιπόν στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι σε όλους καλές διακοπές να δυναμώσετε, να ξεκουραστείτε και να έρθετε με φρέσκι για να ξαναξεκινήσουμε της εργασίας μας. Ευχαριστώ. Καλές διακοπές σε όλους.